συζήτηση με πρώτο σημείο για την κοινή μας συζήτηση την Τραπεζική Ένωση. Εκθέσεις Χακμάρκ, πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση επιστοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων σε περίπτωση κρίσης και την σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Σάιμον συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Έκμαρκ, για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Uh, Κυρία Πρόεδρε, σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε για τα θεμέλια της Τραπεζικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης με την οδηγία για την εξυγίανση των πιστοτικών ιδρυμάτων να είναι η βάση. Πέρσι στις 11 οποίο καταφέραμε να φτάσουμε μια πολιτική συμφωνία για έναν πραγματικά καινοτόμο τρόπο του νομοθετήν. Ω τώρα δεν είχαμε περιθώρια για να δούμε πώ θα χειριστούμε την τραπεζική κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικά ε, επίπεδα. Το νέο αυτό νομοθέτημα ορίζει τι θα συμβεί και τι θα πρέπει να διασώζεται σε περίπτωση κρίση με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο για τους φορολογουμένους και την ε, οικονομική σταθερότητα. Ορίζει την αρχή του bail-in, πράγμα που σημαίνει ότι οι τράπεζες, οι μέτοχοι και οι πιστωτέ θα είναι οι πρώτοι που θα, θα πρέπει να υποστούν τι ζημίε από μια τραπεζική αποτυχία. Και επίση πώ ε, το κράτο ε, υποδοχή και το κράτος εγκατάστασης θα μπορούν να, διαχωρίσουν τις αρμοδιότητές τους. Επίσης, με το νέο νομοθέτημα ορίζεται ότι ενώ το bail-in θα είναι ο βασικός τρόπος για την επίλυση προβλημάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις συστημικών κρίσεων θα χρειάζεται και δημόσια παρέμβαση. Κανείς στο μέλλον δεν θα πρέπει να εικάζει ότι οι φορολογούμενοι είναι εκείνοι που θα διασώζουν τις τράπεζες. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την πιθανότητα ότι θα υπάρχει ανάγκη δημόσια παρέμβαση για να πετύχουμε τη χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα. Και χαίρομαι που εδώ πετύχαμε το σωστό σημείο ισορροπία. Η οδηγία για την ανάκαμψη των τραπεζών ορίζει και τα θεμέλια για την Τραπεζική Ένωση, όπω προείπα, και με τον κοινό μηχανισμό ε, διάσωση. Έτσι, θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνε για όλα τα κράτη-μέλη και θα διέπουν όλη τη λειτουργία όλων των Ιδρυμάτων στην Ένωση. Το βρίσκω καθοριστική σημασία σε αυτό, Πρόεδρε, διότι σημαίνει ότι όταν γίνονται συζητήσει για την Τραπεζική Ένωση πλέον, δεν θα έχουμε μια κατακαιρματισμένη ένωση σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα. Θα υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα τη οποία ακρογωνία λίθο θα είναι η οδηγία ακριβώ αυτή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το σκεφτούμε για το μέλλον, γιατί είναι ο πυρήνα ε, των όσων εξελίξεων θα ακολουθήσουν. Η ευρωπαϊκή οικονομία και οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ θα πρέπει να ε, αντιδρούν με τρόπο ενιαίο και να κινητοποιούμε του κοινού μα πόρου στι διάφορε αγορέ, ώστε να μπορούμε να τι ε, κινητοποιήσουμε σε μια κοινή αγορά. Κυρία Πρόεδρε, κοιτάζοντα και το απότερο μέλλον. Το θέμα είναι τι άλλα, τι θα εξεταστούν στα πλαίσια του οικονομικού τομέα, όχι μόνο σε αυτή τη θητεία αλλά και στι επόμενε. Πράγματα που ίσω δεν τα έχουμε ξαναδεί ω σήμερα. Γι' αυτό θα ήταν μια ευκαιρία τα επόμενα χρόνια να τα χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε το όλο θέμα, να δούμε πόσο προχωρήσαμε, πόσο επιτύχαμε και τι αποτελέσματα θα πετύχουμε αφού εφαρμοστεί όλη αυτή η νομοθεσία. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε Πώ οι ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές θα λειτουργήσουν βάσει αυτών των κανόνων. Με όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια των νομοθετών που έχει γίνει ω τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τώρα θέτουμε τα θεμέλια για, μια σταθερ... για ένα σταθερό τραπεζικό τομέα. Αλλά ταυτόχρονα προσφέρουμε ευκαιρίες για τη λήψη δυναμικών αποφάσεων. Διότι τονίζουμε την ανάγκη υπευθυνοποίηση του της κάθε αρχής διαχείρισης της κάθε τράπεζας. Η τράπεζες και τραπεζίτες δεν μπορούν πλέον να έχουν την αυτοπεποίθηση ή την αίσθηση ότι κάποιος άλλος θα τους διασώσει. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και αίσθηση ευθύνης οι ίδιοι. Και οι επενδυτές βλέπουμε ότι θα πρέπει να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους ε, για να επενδύσουν στον τραπεζικό τομέα ξανά. Στα κεφαλαϊκά επίπεδα έχουμε νέου ναι, νέους κανόνες, νέους για τι τραπεζικέ αγορέ για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τα, για τα παράγωγα προϊόντα και ούτω καθεξή. Όταν τα κοιτάξουμε όλα αυτά, βλέπουμε ότι έχουμε πετύχει πολλά. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε πώ λειτουργούν όλα αυτά στην πράξη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε και κάποια επιμέρου στοιχεία που θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε μια δυναμική χρηματοπιστωτική αγορά είναι πολύ σημαντικό η ευρωπαϊκή οικονομία να ανακάμψει και να ε, αναπτυχθεί. Είμαι υπερήφανος για το αποτέλεσμα του έργου μας. Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους μου για την επικοδομητικότατη συνεργασία και το θετικό πνεύμα εντό του οποίου συνεργαστήκαμε. Ευχαριστώ Ελίζα, Βουλ, Φίλιπ, Βίκη και το τους συνεργάτες σας Ευχαριστώ την γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την ε, εμπειρογνωμοσύνη τους και τι ειδικέ του προσπάθειε και εσά Επίτροπε Μπαρνιέ, για όλο σα το έργο. Έχουμε προλιάνει το έδαφος για έναν τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη που είναι σταθερότερος και να δημιουργήσει νέες θέσει απασχόληση και προοπτικές για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον άλλο μας εισηγητή, τον κύριο Σάιμον, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκείνοι που κάθονται εκεί μπροστά και εργάστηκαν στο φάκελο αυτό, είναι συνοδοιπόροι. Επί πέντε χρόνια, ο, κατά τα οποία εργάστηκε το Κοινοβούλιο για την Τραπεζική Ένωση που ολοκληρώνεται σήμερα έγκαιρα στο τέλος της θητείας μας, έγκαιρα για τους φορολογουμένους, γιατί με την Τραπεζική Ένωση καταφέραμε για πρώτη φορά να βγάλουμε από τη γραμμή πυρός τους φορολογουμένους και να τους βάλουμε στα στις πίσω θέσεις. Δεν είναι πια στην πρώτη γραμμή όταν υπάρχουν τραπεζικές κρίσεις ε, καταφέραμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο ε, μαζί με την εποπτεία τη δημιουργία της ε, αρχής διεκπαιρέωσης να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αντιμετώπισης των κρίσεων, ένα σύστημα διασφαλίσεων το οποίο βεβαίως ε, έπρεπε να προχωρήσει ξεπερνώντας πολλά εμπόδια ε, και μπορούμε να πούμε ότι άξιζε τον κόπο που αφιερώσαμε όλον αυτόν τον χρόνο, άξιζε ε, η πρώτη ανάγνωση και τώρα με την, κλείνουμε την νομοθετική διαδικασία με τη δεύτερη ανάγνωση γιατί καταφέραμε πολλά. δυόμιση-τρία χρόνια πριν δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Το Συμβούλιο δεν θα είχε συμφωνήσει. Ε, αν δούμε το Ταμείο Εγγύης των Καταθέσεων ε, παλαιότερα, το Συμβούλιο είχε συμφωνήσει περίπου στα μισά από αυτά που συμφωνήσαμε τώρα. Έχουμε δηλαδή επιτύχει διπλάσια σταθερότητα για τους φορολογουμένους. Διπλάσια ε, σταθερότητα σε περίπτωση κρίσεων όπου οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν εκείνη ε, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τώρα ε, έγκαιρα ε, διασφαλίσαμε πρόσβαση από την πλευρά του φορολογουμένου του καταθέτη στις καταθέσεις του. Ε, μέσα σε μια εβδομάδα ε, για τον τρεχούμενο λογαριασμό θα μπορεί να εξασφαλίζεται η πρόσβαση. Τώρα έχουμε διευκολύνει τα συστήματα σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε σε πολλά κράτη-μέλη παλαιότερα. Τώρα έχουμε εισαγάγει και στον τραπεζικό τομέα ε, την αρχή ότι θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο οι τράπεζες. Τώρα δηλαδή έχουμε βάλει σε σωστά πλαίσια το σύστημα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλα αυτά πρέπει να καταξιωθούν στην πράξη και βεβαίως αν δούμε λεπτομέρειες θα ε, δούμε ότι υπάρχει και ανάγκη κάποιων βελτιώσεων. Αλλά είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο, σύσσωμο όπως και η Επιτροπή και το Συμβούλιο, στην επόμενη θητεία τους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές. Και θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω για αυτό που πετύχαμε μέχρι τώρα τους σκιώδεις εισηγητές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επικεφαλή στον Επίτροπο Μπαρνιέ και ιδιαίτερα τη Λιθουανική Προεδρία η οποία επέδειξε το θάρρος, την τόλμη να θέσει πάλι στην ημερήσια διάταξη το δύσκολο αυτό φάκελο της ε, εγγύησης των καταθέσεων. Σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και αυτή είναι μια καλή ημέρα για τους πολίτες και τους φορολογουμένους στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στο Συμβούλιο. Ο Υπουργό κ. Βενιζέλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεωρώ μεγάλη τύχη και τιμή το γεγονός ότι εκπροσωπώ το Συμβούλιο σε αυτή τη τόσο σημαντική συνεδρίαση. Μια συνεδρίαση στην οποία γίνεται ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ένωσης. η ταχεία ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στέλνει ένα καθαρό και σαφές μήνυμα σε όλους εκείνους που αμφέβαλαν και την ικανότητα της ευρωπαϊκής ένωσης να αντλήσει τα σωστά διδάγματα από την οικονομική κρίση και να προβεί στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αφορούν την εποπτεία και τη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. η συγκρότηση μιας στέρεης τραπεζικής ένωσης είναι απαραίτητη για την διάρρηξη του δεσμού μεταξύ του τραπεζικού τομέα και του δημόσιου χρέου μεταξύ της δημοσιονομικής και της χρηματοοικονομικής κρίσης που βιώνει η ευρωπαϊκή ένωση τα τελευταία πολλά χρόνια. είναι επίσης ζωτική σημασίας για την αντιμετώπιση του κατακαιρματισμού της αγοράς ιδίως της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της ευρωζώνης. η τραπεζική ένωση έχει συγκροτηθεί σε λιγότερο από δύο χρόνια. πρόκειται για έναν τάνιο άθλο που θα επιτρέψει στην ευρώπη να βγει ισχυρότερη από την κρίση. είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης που θα βασίζεται στην ολοκλήρωση και την αλληλεγγύη στη ζώνη του ευρώ και το ελάχιστο κοινό κανονιστικό πλαίσιο το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί η τραπεζική ένωση προσφέρει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα στο σύνολο της ευρωπαϊκής ένωσης και στην εσωτερική αγορά. ως μέρος αυτού του ελάχιστου κοινού κανονιστικού πλαισίου έχουμε ήδη υιοθετήσει το 2013 χιλιάδες το νομοθετικό πακέτο της οδηγίας τέσσερα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. αυτό εξασφαλίζει τη διατήρηση από όλες τράπεζες επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων και ρευστότητας και ενισχύει την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τον κίνδυνο. με τον τρόπο αυτό ανταποκριθήκαμε και στις διεθνείς δεσμεύσεις της ένωσης στο πλαίσιο της βασιλείας 3. επίσης ως μέρος του ελάχιστου κοινού κανονιστικού πλαισίου οι οδηγία σχετικά με τα συστήματα εγγύηση των καταθέσεων είναι ζωτική σημασίας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνο τη μαζική απόσταση καταθέσεων και να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. έτσι προστατεύονται οι καταθέτε μέσω τη σημαντική ενίσχυση των ταμείων εγγύηση καταθέσεων και μέσα από τη μείωση των καθυστερήσεων στην αποζημίωσή του σε περίπτωση χρεοκοπία των τραπεζών αυτό φυσικά πρέπει να συμπληρωθεί με ειδικότερε διατάξει για την προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του καθώ και των καταθέσεων των μικρών δημόσιων αρχών καθώ και ορισμένων καταθέσεων για στεγαστικού και κοινωνικού σκοπού. προσβλέπω εκ μέρου του συμβουλίου στην επιβεβαίωση από αυτήν την σύνοδο τη ολοκλήρωση τη οδηγία σχετικά με τα συστήματα εγγύηση των καταθέσεων μέσω της έγκρισης της θέσης που συμφωνήσαμε με το κοινοβούλιο στο τέλος του περασμένου έτους. απότερη φιλοδοξία είναι φυσικά να περάσουμε από την οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. ελπίζω ότι αυτό δεν θα αρχίσει να γίνει αντιληπτό ως ζωτική ανάγκη για την ευρωζώνη και την ένωση συνολικά. η οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίαση των τραπεζών είναι επίσης ένα σημαντικό κείμενο υποστηρικτικό της τραπεζικής ένωσης για την οποία ζητείτε σήμερα η έγκρισή σας. η οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίαση των τραπεζών θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες των τραπεζών να ανακάμπτουν μέσα από μια δύσκολη κατάσταση. στην ακραία περίπτωση που μια τράπεζα πλήττεται ανεπανόρθωτα θα επιτρέψει τη διατήρηση των κρίσιμων λειτουργιών της τράπεζας ενώ η εξυγίανση της τράπεζας θα γίνει με συντεταγμένο τρόπο το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τους ιδιοκτήτες και τους ανασφάλιστους πιστωτές όχι τον φορολογούμενο. οι εποπτικές αρχές της τράπεζας και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης θα έχουν πλέον τα μέσα να επιβάλλουν πλήρως αυτή τη διαδικασία. επιτρέψτε μου μια παρατήρηση για τον εποπτικό πυλώνα για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. ο κανονισμός για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό έχει δημιουργήσει μια ισχυρή τραπεζική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ και τα άλλα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα υποπτεύει απευθεία τι συστημικά σημαντικέ τράπεζε και συνεργάζεται πλέον στενά με τι αρμόδιε εθνικέ αρχέ που είναι υπεύθυνε για τι υπόλοιπε. αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και αυστηρότερη εποπτεία του τομέα. τώρα σε σχέση με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανση πρέπει να τονίσω ότι χαιρετίζω εκ μέρου του συμβουλίου θερμά το γεγονό ότι είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε απόλυτη συμφωνία επί του κανονισμού. αυτό θα σας δώσει τώρα τη δυνατότητα να ψηφίσετε για ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα. δεν είναι καθόλου μυστικό ότι η διαδικασία ήταν πολύπλοκη και δύσκολη. πιστεύω ότι ο λεπτός συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε είναι ένα πραγματικό επίτευγμα. όπως συμβαίνει με κάθε συμβιβασμό κανένας δεν τον θεωρεί ιδανικό αλλά το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό για να επιτρέψουμε στην αναζήτησή μας για τελειότητα να υπονομεύσει τη δυνατότητα μιας αποδεκτής συμφωνίας θέσαμε στους εαυτούς μας ένα πολύ φιλόδοξο στόχο είμαστε τώρα πολύ κοντά στο να πετύχουμε αυτό που είχαμε θέσει ως ε, επιδίωξη. έχουμε δημιουργήσει θεμελιώδεις εγγυήσεις για τους φορολογούμενους και τους καταθέτες που θα προστατεύουν τη χρηματοπιστωτική μας σταθερότητα και θα απολαμβάνουν μελλοντικές κρίσεις. θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τους εισηγητές τους σκιώδεις εισηγητές τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής οικονομικών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την μεγάλη του συμβουλή και συμβολή τα επιτελεία του, φυσικά τον επίτροπο κύριο μισελ μπαρνιέ ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά την προηγούμενη προεδρία τη λιθουανική για όσα έκανε και θέλω να διατυπώσω προσωπικά τις ευχαριστίες μου στον έλληνα υπουργό οικονομικών τον κύριο γιάννη στουρνάρα που προεδρεύει την περίοδο αυτή του ecofin στον μόνιμο πρόεδρο του eurogroup καθώς και σε όλους εκείνους που συνέβαλαν άμεσα ή έμεσα σε αυτό το θεσμικό επίτευγμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Και τώρα λόγο στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Όντως είναι μια σημαντική στιγμή η σημερινή και για το κοινοβούλιο σας, αλλά και επειδή με τα τρία αυτά κείμενα τα οποία αποτελούν ένα σύνολο, οικοδομούμε κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές μαζί, μαζί με την Προεδρία, το οικοδόμημα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά βγαίνει από τις δυσκολίες από τις οποίες χτυπήθηκε από το 2008 με μια πολύ βία οικονομική κρίση η οποία κατέστρεψε την ανάπτυξη, αύξησε το δημόσιο χρέος και δημιούργησε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δυσκολίες που συνεχίζουμε σε έναν βαθμό να αντιμετωπίζουμε. Για να αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή, από το Φεβρουάριο του 2010 μαζί, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, μαζί δουλέψαμε, συνεργαστήκαμε και εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη στήριξη του Προέδρου Μπαρόσο σας παρουσίασα 40 σχέδια νομοθετημάτων για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή, να πάρουμε τα μαθήματα που επιβάλλεται να πάρουμε και να οδηγηθούμε σε σταθερότητα. Στο όνομα αυτή τη σταθερότητα, λοιπόν, και ευχαριστώ και τον κύριο Καρά που είναι εδώ, οδηγηθήκαμε σε ένα κεντρικό κείμενο που είναι τα εποπτικά μέτρα για 300 τράπεζες από τις 28 χώρες μέλη. Πήγαμε όμως και πιο μακριά, φτάσαμε σε ένα κώδικα δεοντολογίας με το single book, με τις εγγύσεις καταθέσεων και, τα... και την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίαση τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τους συζητητές, τον κύριο Ζήμον και τον κύριο Χόκμαρκ και όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, την πρόεδρο Σάραν Μπόλς και τους κοιόδους συζητητές. Καταλήξαμε στα δύο αυτά κείμενα τα οποία διέπουν την ενιαία αγορά και καταλήξαμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία με την ενιαία ρύθμιση για τη διαχείριση των κρίσεων με κοινά μέτρα πρόληψης, προετοιμασίας, διαχείρισης και χρηματοδότησης των τραπεζών που αποτυχαίνουν, χωρίς, όπως γινόταν κατά το παρελθόν, να ζητάμε από τον φορολογούμενο τη διάσωση, χωρίς να ζητάμε πια από τον φορολογούμενο να πληρώσει για τις αδυναμίες των τραπεζών το καθήκον μας, που ήταν έτσι κι δύσκολο, έγινε ακόμα πιο δύσκολο εξαιτία της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης. Από το 2010 η δημοσιονομική αυτή κρίση των αγορών συνοδεύτηκε και από κρίση δημοσίου χρέους, ιδιαίτερα οξυμένη κυρίως στην Ευρωζώνη. Συνεπώς έπρεπε να περάσουμε σε μεγαλύτερη ταχύτητα, με μια πιο προθυμένη ολοκλήρωση και με την δημιουργία ε, νέου εποπτικού μηχανισμού που να συνοδεύεται και από τα μέτρα διαχείρισης των κρίσεων. Πρόκειται για την Τραπεζική Ένωση που σας παρουσιάζω από τον Σεπτέμβριο του 2012 σε δύο στάδια. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τις Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κυπριακή, την Ιρλανδική, τη Λιθουανική και βέβαια χαιρετίζω εδώ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, την ελληνική προεδρία δηλαδή που δραστηριοποιήθηκε όλος ιδιαίτερος και την ελληνική κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Στουρνάρα και τους συνεργάτες τους. Περάσαμε λοιπόν σε αυτήν την μεγαλύτερη ταχύτητα και την φιλοδοξία μας την συμμερίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή και από πριν ακόμα. Από το 2010 η Ελίζα Φερέιρα ε, είχαμε τη δικιά σας νομοθετική έκθεση που υπενθύμιζε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο την διαχείριση της τραπεζικής κρίσης και ζητούσε ένα ταμείο σταθερότητας. Με μια ενότητα καταλήξατε στο ψήφισμά σας, το οποίο τελικά έγινε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλέψαμε. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια προσέγγιση ρεαλιστική Περάσαμε το πρώτο στάδιο με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που είναι πιο αυστηρός για όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης και που ισχύουν πια οι ίδιοι κανόνες για όλες τις τράπεζες. Οι κανόνες της ενιαίας αγοράς με αυτό τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Με πιο ομοσπονδιακή και πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Χαιρετίζω εδώ το έργο της Μαρίας Τίεσεν και όλων των σκιωδών εισηγητών. Χαιρετίζω επίσης και τη δουλειά που έγινε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον Λουί, τον αντιπρόεδρο της Αμπίνα Σλέτιγεν που δούλεψαν σκληρά για τον μηχανισμό αυτόν τον εποπτικό που ουσιαστικά λειτουργεί ήδη για τις δοκιμές αντοχής που θα έχουν σαν αποτέλεσμα αν υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Η Τραπεζική Ένωση όμως πρέπει να στηρίζεται στα δυο της πόδια. Υπάρχει η εποπτεία, υπάρχει και η εξυγίαση. Δεν ήταν εύκολο και ήταν ίσως πιο δύσκολο να καταλήξουμε στην εξυγίανση από ότι στην εποπτεία. Και αυτό γιατί εδώ διακυδεύονται σημαντικά πράγματα και οι αρχικές θέσεις ήταν πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους. Επιδείξατε ρεαλισμό όμως χρειάστηκε προσπάθειες για να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό και η συμφωνία τη 20 η Μαρτίου αποτελεί μια τεράστια πρόοδο. Γι' αυτό και ευχαριστώ ένθερμα την Ελίζα Φερέιρα και την πρόεδρο Σάραν Μπόλ και την ε, κυρία Βόρτμαν Κόλ που είναι εδώ, τον Σβέν Κιγόλ, τον Βίκη Φόρτ που δούλεψαν σκληρά καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που κράτησαν μερικές φορές 17 ώρες για να καταλήξουμε στη συμφωνία αυτή. Πιστεύω ότι σοβαρά φέραμε σε πέρα στην αποστολή μας. Θέσαμε τις προϋποθέσεις ώστε οι τραπεζές μας να είναι πιο ισχυρές στο τραπεζικό μας σύστημα και η εμπιστοσύνη στο ευρώ και στις τράπεζές μας να ανακτηθεί. Πολύ σύντομα για αυτούς που μας παρακολουθούν εκτός κοινοβουλίου πρέπει να πω ότι έχουμε αλλάξει πράγματα. Από εδώ και πέρα θα είναι οι μέτοχοι και οι που θα χρηματοδοτούν την αποτυχία μιας τράπεζας μέσω διάσωσης με ίδια μέσα και υπάρχει και το σύστημα αυτοεγγύσεων καταθέσεων που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Είναι σύστημα το οποίο άρχισε να ισχύει πριν από 5-6 χρόνια ουσιαστικά. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι ότι ο αριθμός των τραπεζικών ε, κρίσεων όπου χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν χρήματα από το φορολογούμενο ε, μετρείται στα δάχτυλα του νοσχεριού. Δεύτερο σημείο. Προστασία των καταθετών. Πρέπει να επιβεβαιωθεί και πάλι κάτω από 100.000 ευρώ, πάντα παντού, κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις υπάρχει εγγύηση των καταθέσεων αυτών και ο κίνδυνος απώλειας είναι πολύ αδύναμος εξαιτία της ρύθμισης αυτής προστασίας των ε, μικρών καταθετών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έπειτα στο σύνολο της Ένωσης προβλέπουμε προετοιμασία για τις κρίσεις. Σε δημοσιονομικά ζητήματα βλέπετε, όπως και όταν έχουμε οικολογικές καταστροφές που πολλαπλασιάζονται, η πρόληψη τελικά στοιχίζει λιγότερο από τη θεραπεία από την αντιμετώπιση δηλαδή των κρίσεων. Όταν πρέπει να αντιμετωπιστεί μια κρίση η οποία έχει λάβει χώρα, ξέρουμε ότι αν έχουμε προετοιμαστεί, χρειάζεται να ξοδέψουμε λιγότερα από ότι όταν περάσουμε σε ασύνταχτη αντιμετώπιση της όποιας κρίσης. Αυτό ισχύει και στις τράπεζες. Στο μέλλον λοιπόν η κάθε τράπεζα πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί να διασωθεί χωρίς να κινδυνεύει να πλήξει την οικονομική σταθερότητα τέρμα πια στους αυτοσχεδιασμούς. Τέταρτον, στην Ευρωζώνη και σε όλες τις χώρες μέλη που θέλουν να συμμετέχουν στον μηχανισμό αυτό, υπάρχουν ενίοι κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν για όλες τις τράπεζες. Υπάρχει το Συμβούλιο Εξυγίανσης με έναν μηχανισμό ευρωπαϊκό εξυγίανσης. Υπάρχει ένα σύστημα αξιόπιστο, περίπλοκο. Εντάξει, και εγώ λυπάμαι γι' αυτό. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσπαθούν να δούνε τι θα γίνει με τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Πάντως, οι ευθύνε που αναλαμβάνει το Συμβούλιο αυτό είναι τεράστιες. Το σύστημα βασίζεται σε μια αξιόπιστη χρηματοδότηση, επιταχυνόμενη για διάστημα 8 ετών, με την αμοιβεποίηση των συνεισφορών σε επίπεδο 60% και αυτό το οποίο με νοιάζει πολύ είναι η συνοχή της εσωτερικής αγοράς και σας βέβαια. Διατηρήθηκε διότι σεβόμαστε πλήρως την οδηγία για την εξυγίανση που ισχύει στις 28 χώρες μέλη. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, έπρεπε να σας ευχαριστήσω. Εισακούστηκε το μήνυμά σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δούλεψε με φοβερή θέληση και επιμονή. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω εκτός από εσά και τις δικές μου υπηρεσίες και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνεργάστηκαν πολύ καλά μαζί σας. Δεχτήκατε συμβιβασμούς. Δεν ήταν εύκολο. Για παράδειγμα όσον αφορά τη διακυβερνητική συμφωνία, ακόμα και να είναι περιορισμένη, ήταν ε, δύσκολο σε πολλούς από εμά να γίνει δεκτή, αλλά η αμοιβεποίηση της χρηματοδότησης, το Συμβούλιο αυτό της εξυγίανσης, η σταθερότητα των οικονομικών, ο περιορισμός της προθεσμίας για την αποζημίωση των καταθετών, όλα αυτά και πολλά άλλα έγιναν δυνατά χάρη σε εσά, χάρη τη δικιά σας αποφασιστικότητα να διατηρηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας και αξιοπιστίας του κειμένου αυτού. Με την Τραπεζική Ένωση λοιπόν που βασίζεται στα δυο της πόδια, στους δυο της ε, πυλώνες, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια της Ευρώπης μετά το ευρώ. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα δημοσιονομικά κείμενα και εδώ πρέπει να προσέξουμε και τώρα και αργότερα να βλέπουμε τι κάνουν και εταίροι μας στο G20 και όπως είπατε και πριν να φροντίσουμε όντως να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Πρέπει να αφήσουμε δηλαδή κάποιο χρόνο εφαρμογής του συστήματος, να γίνει αξιολόγηση και πιστεύω ότι έτσι όπως δουλέψαμε θα πετύχουμε την σταθερότητα του συστήματός μας. Όπως είπατε και πριν, τώρα που έχουμε την ανάκαμψη, να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η διαφάνεια θα διατηρηθεί, η υπευθυνότητα, όπως είπε και ο κύριος Σίμων, και όντω χρειάζεται και λίγη ηθική εδώ που χάθηκε για ένα διάστημα. Και από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη και την απασχόληση και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο λόγο στου αγορητέ εκπληρωμάτων των πολιτικών ομάδων. Για το ΕΛΚ, πάλι δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Τραπεζική Ένωση θεωρώ ότι είναι λεπτό εγχείρημα στο χρηματοπιστωτικό τομέα αυτής της θητείας και ευχαριστώ και τον, κύριο, τον Επίτροπο Μπαρνιέ και συμφωνώ με τα επιχειρήματά του. Ως κοιόδης ε, του Λαϊκού Κόμματος ε, ήμουν ε, ε, υπεύθυνος ε, και ασχολήθηκα ιδιαίτερα για τον τρίτο πυλώνα της διασφάλισης των καταθέσεων και χαίρομαι που το σημαντικό αυτό θέμα της εγγύησης των καταθέσεων ολοκληρώθηκε και πιστεύω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Το Φεβρουάριο του 2012 στην Ολομέλεια σε πρώτη ανάγνωση παρουσιάσαμε τη θέση μας ε, μετά το μπλοκάρισμα των διαπραγματεύσεων ε, από το Συμβούλιο. Το περασμένο φθινόπωρο, επί Λιθουανικής Προεδρίας, ξανάρχισαν οι διαπραγματεύσεις και μετά από τρεις τριμερείς διαλόγους, ε, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013 βρέθηκε συμφωνία. Υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα τώρα για την διασφάλιση των καταθέσεων. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα. Ε, σημαίνει ότι κάθε καταθέτης μπορεί να έχει εξασφαλισμένες καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ ε, χωρίς ε, άλλες προϋποθέσεις. Έτσι δίνεται προτεραιότητα στους μικροκαταθέτες και αποταμιευτές. Είναι υψηλό το επίπεδο ασφάλειας των καταθετών. Και τώρα υπάρχει και ε, σε ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα ε, αντιμετώπισης των τραπεζών. Με τη σημερινή ψηφοφορία για τους άλλους δύο πυλώνες Τραπεζικής Ένωσης με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και ε, την εγγύηση των καταθέσεων θα έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο θα έχει κάνει ένα βήμα μπροστά πολύ σημαντικό. Η ε, Τραπεζική ε, ε, Ένωση είναι ένα έργο το οποίο καταφέραμε στα πλαίσια αυτής της θητείας να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Θερέιρα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή την ολομέλεια, την τελευταία αυτή τη θητεία, το Ευρωκοινοβούλιο θα εγκρίνει τρία ακόμα νομοθετήματα που είναι θεμελιώδη για την αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων. Ίσως αυτή είναι η σημαντικότερη θητεία μετά την κρίση του 2008, διότι καταφέραμε να διασώσουμε ε, τις τράπεζες και το 20% του ΑΕΠ τέσσερις κοινωτικούς προπολογισμούς και να διασώσουμε επιχειρήσεις και πολίτες από μια κρίση που ακόμη συνεχίζεται. Δεν παραμείναμε αδιάφοροι και μάλιστα το 2010 με την έκθεση που ο Επίτροπος Μπαρνιέ είχε την ευγένεια να ανακαλέσει. Ήδη τότε το Ευρωκοινοβούλιο πίεζε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με τόλμη και διορατικότητα. Και χάρη ακριβώς στη δράση του Επιτρόπου Μπαρνιέ και της ομάδας του ήρθε η απόκριση. Οι τράπεζες έχουν πλέον προστατευθεί. Έχουμε διασώσει την ε, υγεία των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και οικογενειών. Τώρα πλέον μπορούμε τις τραπεζικές κρίσεις να τις, αντιμετωπίσουμε προκαταβολικά, να προβλέψουμε τη διάσωση με ίδια μέσα για να προστατεύσουμε καταθέτες και επιχειρήσεις και τράπεζες, να αντιμετωπίσουμε τον κάθε κίνδυνο και να έχουμε και εθνική εγγύηση για τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Για την Ευρωζώνη και τις, τα μέλη της είναι μεγαλύτερες οι φιλοδοξίες. Έχουμε ενιαίο μηχανισμό επιπτίας ε, που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ισχυρή ε, εποπτεία με ένα εύρωστο τραπεζικό σύστημα. Αυτό ακριβώς θα εγκρίνουμε σήμερα. Ως εισηγήτρια είμαι πεπισμένη και θα επιβεβαιωθεί πιστεύω εδώ ότι μπορεί η συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου να βελτιώσει ιδιαίτερο το κείμενο του Συμβουλίου. Το καθεστώς που προβλέπουμε θα μπορέσει να μας προστατεύσει από αφαιρεγγιότητες, περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας τραπεζών και να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις από τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα κοινό εργαλείο εξυγίανσης με μία προβολή σε μία τριετία ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η παρέμβασή μας. Επειδή η τριγμή ήταν πολύ σοβαρή ως τώρα, ε, γι' αυτό και οι δικές μας δεσμεύσεις είναι τελείως ειλικρινείς. Να ευχαριστήσω την Σάρον, την, Σάρον, την Κορίν, τη Σιλβή, ε, τις γυναίκες και τους άντρες που συμμετείχαν στη δημοτευτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για την ε, δέσμευση και την ε, ανθεκτικότητά τους αλλά και τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων που επέτρεψαν ήδη στη δική μου την ομάδα, του σοσιαλιστέ και δημοκράτες να προχωρήσουμε. Αλλά και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Στάθηκαν στο πλευρό μας και επέτρεψαν την πολιτική ε, υλοποίηση των πεπιθήσεών μας. Από κοινού μπορέσαμε την διαπραγμάτευση αυτή να την οδηγήσουμε σε επιτυχία με πυγμή και με ε, αποφασιστικότητα. Το Συμβούλιο το κατάλαβε αυτό και ευχαριστώ την Ελληνική Προεδρία και τον Υπουργό ε, Γιάννη Τουρνάρα αλλά και τον κύριο Ντίσεμπλουμ για τις ε, δυνατότητες στη διαπραγμάτευση να βρούμε θέσεις σύγκλησης Αλλά και όλη την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διευκόλυναν τη σύγκληση αυτής της απόψης. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας, διότι χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Γι' αυτό χαιρετίζουμε και τη συμβαστική πρόταση του Συμβουλίου υπό την έννοια ότι η κύρωση της διακυβερνητικής συμφωνίας από τις 2 Ιανουαρίου 2016 θα διασφαλίσει μια γραμμή πιστώσεων που θα μπορέσει να λειτουργεί από τη θέση σε ισχύ ε, της ε, οδηγίας αυτής για το Ταμείο Εξυγίανσης. Η προληπτική κεφαλαιοποίηση είναι μία αρχή που θα επιτρέψει να μην, φορολογ... χρηματοδοτούν πλέον οι φορολογούμενοι της τράπεζας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο τρίτο πυλώνα τη Τραπεζική Ένωση είναι το ενιαίο σύστημα τη εγγύηση των καταθέσεων που τώρα έλειπε. Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν έχει θέσει τα θεμέλια για να πάυσει η τάση των τραπεζών και των κρατών να εξασφαλίζουν μέσω των καταθέσεων των φορολογουμένων ε, την διάσωση τραπεζών και επιχειρήσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο επιτέλους διασφαλίζει και ελπίζουμε να το συνεχιστεί αυτό στη φάση της υλοποίησης να μην χαθούν όσα πετύχαμε με τόσο κόπο. Ευχαριστώ όλου. Ευχαριστούμε για την άλλη ο κύριος Κλίντς για λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Επικριθήκαμε ότι ε, προκαλέσαμε ένα τσουνάμι με τις ρυθμίσεις μας που εγώ όμως νομίζω ότι όλες ήταν σωστές και απαραίτητες ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην ασφάλεια του τομέα αυτού. Είπε και ο Επίτροπος Μπαρνιέ ότι είχαμε θέσει λάθος προτεραιότητες. Έπρεπε να αρχίσουμε πρώτα με την Τραπεζική Ένωση, ε, η οποία στόχο έχει να ε, σταματήσει αυτή την ε, υπερβολική και ασφιχτική διασύνδεση μεταξύ τραπεζών και κρατών κυβερνήσεων. τώρα δεν έχουμε πια ρυθμιστικό αρμπιτράζ, έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών. Ο φόβος ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ε, νομισματικής πολιτικής ε, και ε, οικονομικής πολιτικής νομίζω ότι ο φόβος αυτός δεν είναι ανυπόστατος και ε, δεν διακινδυνεύει, δεν υπονομεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τον μηχανισμό ε, πρακτικής διεκπαιρέωσης, νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξυγίανσης χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Θα υπάρχει δυνατότητα ε, κάλυψης ε, των φορολογουμένων και των καταθετών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που είχαμε κατά νου κοινοβούλιο, αλλά είναι αποδεκτό. 8 χρόνια και όχι 10 για τη χρηματοδότηση, ε, μέχρι δύο χρόνια στο 60% ε, ε, όμως είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή θα πρέπει οι μικρές τράπεζες και τα ταμιευτήρια ε, να αντιμετωπιστούν με την αρχή της αναλογικότητας και να μην ε, υπερτιμάται και να υπολογίζεται σωστά ο κίνδυνος κάθε πιστοτικού ιδρύματος. Νομίζω ε, και έχω εμπιστοσύνη στον, και στον Υπουργό κύριο Βενιζέλο ότι θα προχωρήσουμε στην ταχεία εφαρμογή όλων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λάμπερτ για τους πράσινους. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποτέ πια. Πόσες φορές δεν ακούσαμε αυτά τα λόγια. Ποτέ πια ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να διασώνει μια αποτυχημένη τράπεζα. Ποτέ πια. Σήμερα μόνο, στη τελευταία θητεία, στη τελευταία μάλλον σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της θητείας αυτής, γίνεται πραγματικότητα η φιλοδοξία αυτή να προστατεύσουμε το φορολογούμενο από τι αποτυχίε του τραπεζικού τομέα. Το κείμενο, το οποίο, τα κείμενα μάλλον που θα εγκριθούν σήμερα αποτελούν πρόοδο, αναμφισβήτητα, σαφέστατα. Οι μέτοχοι, οι πιστωτέ των τραπεζών είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνουν πολύ πριν από το φορολογούμενο. Όμω, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα κράτη-μέλη, και αυτό με εξέπληξε, με τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη στήριξη μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω των υπηρεσιών του κυρίου Ρεν, που είναι φιλελεύθερο αγωνίστηκαν για να συμπεριλάβουν και τη ρήτρα προληπτικής ανακεφαλοποίησης που επιτρέπουν στις χώρες να βοηθούν τις τράπεζες πριν φτάσουν σε αποτυχία. Δηλαδή, αν οι αγορές δεν εμπιστεύονται μία τράπεζα, τότε τα κράτη να τις βοηθούν. Εμένα με εκπλήσει η αντιμετώπιση αυτή, γιατί, αυτός, γιατί νόμιζα ότι θα λέγαμε ότι η ανακεφαλοποίηση θα γίνεται μόνο αν γίνει έγκαιρα από πριν. Είναι απαράδεκτο λοιπόν αυτό. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν τράπεζες να είναι ε, διακρατικές ε, όταν ζουν και να γίνονται εθνικές όταν αποτυχαίνουν. Ο ενίο επαγγελματικό μηχανισμό αποτελεί μια πρόοδο δεδομένου ότι πηγαίνουμε σε μια μεγαλύτερη ομοσπονδιοποίηση της διαχείρισης κρίση. Αλλά και πάλι οι μεγάλε τράπεζε όταν θα αντιμετωπίζουν δυσκολίε, θα διαχειρίζονται από ένα συμβούλιο του κράτου και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο, κύριε Μπαρνιέ, αυτό που με θλίβει σε σχέση με τη δικιά σα δράση είναι ότι το αρχικό κείμενο το οποίο θα έπρεπε να βάλει ένα τέλος ε, στις ε, κακές τράπεζες φτάνει πολύ αργά με τέτοιο τρόπο που η θητή αυτή, αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να χειριστεί αυτό το θέμα. Οι τράπεζες που θεωρούνται πολύ μεγάλες για να αποτύχουν, για να τις αφήσουμε να αποτύχουν, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Το κείμενο το οποίο εσείς υποβάλλατε πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε αυτή τη φορά να το επεξεργαστούμε και να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για τους και μεταρρυθμιστές, κυρία Φόρτ, δύο λεπτά. Σήμερα ε, εξετάζομαι τρία μέρη. Το πρώτο είναι η παγκόσμια αλλαγή που αφορά τα λάθη του παρελθόντος. Όταν αντιμετώπιζαν ε, αποτυχίες οι τράπεζες θα έπρεπε ε, ή να προχωρήσουν σε πτώχευση ή σε διάσωση με ίδια μέσα. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Μπορούμε να έχουμε εκαθάριση, ε, τακτική και οι καταθέτες θα μπορούν να προστατεύονται. Ο χρηματοοικονομικός κόσμος θα είναι ασφαλέστερος. Χάρη στο έργο και του G20 ε, τη, ε, τώρα ε, έχει ε, εγκριθεί ένα κομμάτι ε, πολύ σημαντικό από την παγκόσμια πρακτική. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εγγύηση των καταθέσεων. Βεβαίως δεν θα πρέπει οι καταθέτες να πληρώνουν τον λογαριασμό. υπάρχουν σε ορισμένες χώρες ταμεία προστασίας καταθέσεων. Άλλες χώρες όπως η δική μου εισέπραξαν μια εισφορά, ένα τέλος για τη δημιουργία δομών προστασίας. Ε, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν χρειάζεται μια συνταγή για όλους και καλό είναι που το σεβαστήκαμε αυτό. Το τρίτο πυλώνα είναι η Τραπεζική Ένωση. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να κάνει ένα βήμα παραπέρα και οι αποφάσεις που ελαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών τώρα θα λαμβάνονται περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συνένωση κονδυλίων και κεφαλαίων. Λόγω της Ευρωζώνης ε, ήθελαν κάποιες χώρες μέλη να το κάνουν αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες δεν είναι στην Ευρωζώνη όμως και χαίρομαι που η διακυβερνητική ξεκαθαρίζει ότι δεν μοιραζόμεθα τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Ε, της Ευρωζώνης. Ε, αυτό είναι σωστό για αυτούς που επιλέγουν να μην συμμετάσχουν. Ε, έχουμε μπροστά μας σκληρές διαπραγματεύσεις για να έχουμε τις συμφωνίες που χρειάζονται. Χρειάζονται διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις και κάποιες χώρες καταλαβαίνουν ότι θέλουν πιο εξελιγμένη ευρωζώνη, άλλες όχι. Θα μπορούμε να προχωρήσουμε και για τις δύο. Ευχαριστούμε για την κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ε, προέκυψε η οικονομική κρίση, η ευρωπαϊκή και η διεθνή στριγμή ε, δεν ε, οδήγησαν μάλλον σε μια σειρά από δηλώσεις από όλε τι πλευρέ, με προειδοποίηση ότι θα υπήρχαν δρακόντια μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση και να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Έξι χρόνια μετά και αφού έχουμε επενδύσει το 26% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, δηλαδή τέσσερι κοινοτικού προπολογισμού για να διασώσουμε τι τράπεζε. τελικά αυτό που έγινε έγινε, αλλά με βήματα και ρυθμού χελώνα δυστυχώ, χωρί να πετύχουμε αυτό που θέλαμε η νέα τάξη που δημιουργείται δεν έχει υπερατωθεί και η κρίση δεν έχει τελειώσει. Το εγχείρημα της Τραπεζικής Ένωσης κατά την ε, αντίληψή μου είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της αποτυχημένης ε, υπόσχεσης που δόθηκε. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα σύστημα για τη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών αλλά ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκ των υστέρων θέλησαν να βάλουν σε κεντρικό ρόλο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία ουσιαστικά επιτρέπει την τραπεζική εποπτεία με ανάληψη οποιασδήποτε ε, αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να θελήσει να αναλάβει. Ουσιαστικά είναι η το μη δημοκρατικό θεσμικό όργανο που είναι το πιο ισχυρό στον κόσμο αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τελικά έχει δημιουργηθεί με, αυτή την, ε, με αυτόν τον τρόπο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης μετά από 8 χρόνια όμως τα πάντα μπορεί να συμβούν με αυτή την προοπτική που έχει δοθεί πολλοί μπορεί να αλλάξουν άποψη. Δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτή την υπόσχεση θα τη δούμε λαμβάνει σάρκα και οστά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα με αυτή την δέσμη μέτρων. Διότι αρχίζει να γίνεται αφόρητο το πώς οι μεταρρυθμίσεις επιβάλλονται στην Ευρωζώνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βιώσιμα ε, προγράμματα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά σκοπό έχουν να προστατεύσουν την εσωτερική αγορά από τις οποιασδήποτε διακυμάνσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η κυρία Σενκλέρ. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Πάσκα για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, Πρώτα κύριε Επίτροπε, Στη χώρα μου ο τραπεζικός τομέας είναι υγιής και σταθερός. Με την Τραπεζική Ένωση όμως μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. Ο τραπεζικός τομέας θα κυριαρχείται από το γεγονός ότι θα παρεμβαίνουν τα κράτη. Οι ανεξάρτητοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί τελικά θα αποτελέσουν στόχο για καθάριση από τη χώρα όπου θα υπάρχουν οι μητρικές εταιρείες. Τέτοιες ε, μετατροπές θα πρέπει να αποφευχθούν όπως επίσης και οι μεταφορές ρευτότητας προς το εξωτερικό. Κύριε Επίτροπε, εγώ δεν λέω ότι η Τραπεζική Ένωση έχει μια κρυφή ατζέντα για να καταστρέψει οι υγιείς ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για να προσφέρει ρευστότητα στις μη σταθερές χώρες. Όμως η ίδια διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να υπάρξει μια τέτοια διαδρομή με σημαντικές συνέπειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Συγκλέρα. Δεν είναι όμως εδώ, οπότε ο λόγος στους υπόλοιπους εισηγητές η κυρία Βόρτμαν Κόλλη. για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Σήμερα είναι μια ιστορική σημασία μέρα για την ιστορία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η συμφωνία για τις αρχές τραπεζικής εξυγίανσης είναι το τελικό παζλ, το τελικό κομματάκι του παζλ για την Τραπεζική Ένωση είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό για την ανάκτηση εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό επίση για τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι τράπεζε για την οικονομία μα. Η στάση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο ήταν ζωτική σημασία. Με την ε, απόφαση αυτή τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα και η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε καλή εφαρμογή των κανόνων για την αναδιάρθρωση των ε, προβληματικών τραπεζών. Με τη συμφωνία αυτή καταφέρνουμε να μην πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος, αλλά οι μέτοχοι και οι πιστωτές, οι επενδυτές για τις αποτυχίες των τραπεζών στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, αλλά και στη Γαλλία και στις γερμανικές τράπεζες ακόμα. Οι μέτοχοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στη υπεύθυνη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω και τους συναδέρφους και τον Μισελ Μπαρνιέ και την Προεδρία και τον κύριο Ντάιζενμπλουμ. Να τους ευχαριστήσω όλους που έγινε εφικτή η συμφωνία αυτή. Πρόεδρε, είναι τελευταία φορά που μιλάω εδώ ως Ευρωβουλευτής και ως ε, εκπρόσωπος της ομάδας μου. Είμαι περήφανη για αυτό που πετύχαμε για να αντιμετωπίσουμε την τραπεζική κρίση. Η οικονομική διαχείριση, το six-pack, το two-pack, η δημοσιονομική πολιτική. Όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη. Σήμερα πετυχαίνουμε και την Τραπεζική Ένωση. Είμαστε στο σωστό δρόμο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο ευρώ. Η ανάκαμψη της οικονομίας μας επίσης προχωράει, αλλά μένει ακόμα πολλής δρόμος. Χρειάζεται χρόνος, αλλά και εδώ προχωράμε καλά. Και τέλος, στην Ευρώπη και στις χώρες μέλη πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Είναι πολύ βασικό αυτό για την κοινωνία μας γιατί έτσι θα υπάρξει ανάκαμψη και της εμπιστοσύνης και θα βρεθεί και πάλι απασχόληση για τους πολίτες μας και την νεολαία μας. Περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάντσες Πρεσέντο. Για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά την θητεία μας έχουμε υιοθετήσει σημαντικά νομοθετήματα για θέματα κεφαλαίου και για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δημοσιονομικής Εποπτείας, για να ξεπεραστεί η κρίση, για να υπάρξουν επιστώσεις, για να υποφεληθούμε από τα θετικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Η έγκριση σήμερα των κειμένων αυτών για την εγγύηση καταθέσεων και για ένα κοινοτικό πλαίσιο όσον αφορά την εξυγίανση δημοσιονομικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Θέλουμε να προσφέρουμε ασφάλεια στους καταθέτες και να τους προστατεύσουμε απέναντι σε αποτυχίες τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ βασικό, μια προπόθεση για την επιτυχία τη Τραπική Ένωση και να σταματήσει πια αυτό ο φαύλο κύκλο ε, δημοσίου και ιδιωτικού χρέου, να πάψει πια το πρόβλημα ρευστότητα και πιστώσεων και να προχωρήσει η νομισματική μα πολιτική. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί μετά τον ενίο παπτικό μηχανισμό καταφέραμε ευτυχώ σήμα τσίμα να πετύχουμε και συμφωνία για τα σημερινά κείμενα που σημαίνει αποτελεσματική αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και ένα ενίο μηχανισμό εποπτείας, όμως Συγχρόνως πρέπει να πω ότι η διαδικασία ενίσχυσης του δημοσιονομικού συστήματος πρέπει να συνεχιστεί με διαρθρωτικές αλλαγές και με βελτίωση της Τραπεζικής Ένωσης με έναν νέο μηχανισμό ασφάλειας καταθέσεων και με ένα κοινό δίκτυο. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας γιατί τελικά η Τραπεζική Ένωση απαιτεί και οικονομική και δημοσιονομική ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σμίτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Τραπεζική Ένωση είναι η σημαντικότερη ψηφοφορία που έχουμε, στην οποία έχουμε προχωρήσει σε όλη μας την κοινοβουλευτική θητεία, πιστεύω. Διότι δημιουργεί μια ισχυρή, ένα ισχυρό σύστημα εποπτείας ε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το σύστημα εγγύηση των καταθέσεων και έναν τρόπο να μην χρηματοδοτούν τις τράπεζες οι φορολογούμενοι. Η νομισματική ένωση ευθύ εξ αρχής υπήρξε ένας σημαντικός παράγοντας. Θα έπρεπε να μας βοηθά να ξεπερνούμε την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης. Υπήρξαν τόσες, τόσοι φόβοι ότι θα καταρρεύσει η Ευρωζώνη, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να φύγει από την Ευρωζώνη. Όχι. Είδαμε τώρα πόσο αποφασιστική δράση μπορεί να έχουν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε στιγμές κρίσης. Ήδη το είχαμε ε, το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε στις εθνικές ε, αγορές πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η δράση ε, σε σχέση με πράγματα που είχαν συμβεί τη δεκαετία του 20 και του 30 με το οικονομικό κράχ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έδειξε τη δύναμή τη σε δύσκολε στιγμέ. Η Τραπεζική Ένωση δημιουργεί την απαραίτητη σταθερότητα. Αλλά οι μεταρρυθμίσει πρέπει να συνεχίσουν με αμύωτο ρυθμό. Νομίζω ότι είναι κρίμα που δεν συμμετέχει η Τραπεζική Ένωση, Πρόεδρε, η Σουηδία. Πιστεύω ότι για τι μεγάλε τράπεζε, του ομίλου, του πελάτε του θα ήταν σημαντικό. Και δεν νομίζω ότι θα μα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτό. Είναι η τελευταία μου ομιλία ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Επίτροπο και την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πραγματικά νομίζω ήταν εξαιρετική η δουλειά σα και ελπίζω η χώρα μου κάποια στιγμή να συμμετάσχει στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκίγκολ, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, αγαπητή Προεδρία του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, η Τραπεζική Ένωση είναι το μεγαλύτερο βήμα μπροστά της Ένωσης σε αυτή τη θητεία. Κάναμε αυστηρότερους κανόνες, έχουμε κοινή ευρωπαϊκή εποπτεία και κοινούς ε, κανόνες ε, αντιμετώπισης ώστε στο μέλλον να μην πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι αλλά να αναλαμβάνουν ε, ευθύνη ή ε, υπεύθυνοι στην τραπεζική αγορά. Όμως λείπουν δύο στοιχεία ακόμη, το θέμα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, γιατί ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή και δεν βρήκαμε και λύση για το πρόβλημα των πολύ μεγάλων τραπεζών που ακόμα και με την καλύτερη αρχιτεκτονική ε, θα είναι δύσκολη η εξυγίανσή τους. Ε, γι' αυτό υπάρχει ε, η πρόταση σημαντική από την Κομισιόν που πρέπει να τη συζητήσουμε για τον διαχωρισμό των ε, τραπεζικών εργασιών και των κατηγοριών τραπεζών. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου ποιος ήταν. Σε όλα αυτά τα νομοθετήματα ε, το Κοινοβούλιο ε, επίεσε προς ένα πιο δημοκρατικό, πιο αποτελεσματικό ε, μοντέλο. Επιτύχαμε μεγάλες πρόοδους και γι' αυτό θα ψηφίσουμε και την σχετική έκθεση. Η, παράλληλα όμως θα πρέπει και η ε, διακυβερνητική συμφωνία να ε, προωθηθεί θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές φορές ε, το Συμβούλιο παραβίασε τις αρχές μας χωρίς να εμποδιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τώρα έχουμε το 27.2 το περίφημο άρθρο για την ε, ανακεφαλαίωση των τραπεζών το περιορίσαμε ε, όσο μπορούσαμε. Τώρα όμως βλέπουμε ότι ε, υπάρχει προσπάθεια επανεισαγωγής του από την πίσω πόρτα. Θα πρέπει να ισχύει όμως η ανάληψη ευθύνης και σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε ο κύριος Στρέτσεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, κύριε Επιτροπέ. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι οι τράπεζες θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες, διότι εδώ και χρόνια δανείζονταν χρήματα από τα κράτη, αντί να ε, στηρίζονται στη δική τους, στους δικούς τους πόρους. Και πολλές φορές τα δημόσια ταμεία χρησιμοποιήθηκαν για να διασωθούν οι τράπεζες. Το αποτέλεσμα ως αναμενόταν ε, και ως το αναμενόμενο ήταν μια απόλυτη κατάρρευση. Και δικαίως, διότι η Τραπεζική Ένωση επιτέλους θα πρέπει να επιτρέψει να διαχωρίσουμε το χρέος των τραπεζών από το κρατικό χρέος. Ως τώρα αυτό ήταν ανέφικτο. Και βεβαίω είναι ακόμη δύσκολο, διότι η πρόταση που συζητούμε για την Τραπεζική Ένωση δεν θα κάνει τα κράτη-μέλη να συμπεριφέρονται καλύτερα ή με πιο ε, συμφέροντα τρόπο. Δεν θα μεταρρυθμίσουν ε, ευθύ αμέσω όσα είναι αδύνατο να μεταρρυθμιστούν. Η Τραπεζική Ένωση δεν είναι η σωστή επιλογή, ούτω ή άλλω. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χούντης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πριν από έξι χρόνια είδαμε να καταραίει το χρηματοπιστωτικό σύστημα καζίνο που δημιουργούσε υπερκέρδη για τους πολλούς και τους ισχυρούς ένα σύστημα που έλαβε σε κεφάλαια εγγυήσεις και άλλα δώρα από τα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης περίπου τέσσερα τρισεκατομμύρια ευρώ την ίδια στιγμή που οι άνεργοι στην ευρώπη είναι 26 εκατομμύρια. είδαμε τους προστάτες αυτού του συστήματος τη μαφία των κερδοσκόπων τους οίκους αξιολόγησης να σφυροκοπούν την ελλάδα και να την οδηγούν σε κρίση χρέους και στα μνημόνια και στη συνέχεια να επιτίθεται στην ιρλανδία στην πορτογαλία στην ισπανία στην ιταλία και τέλος στην κύπρο. είδαμε αγαπητοί συνάδελφοι πριν τέσσερα χρόνια την ευρωπαϊκή ένωση την κυρία μέρκελ τον κύριο σαρκοζή τον κύριο παρόζο να θυσιάζουν την ελλάδα ώστε να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως με περισσή κοινικότητα μας ομολόγησε ο κύριος όλι Ρεν. κυρία πρόεδρε η τραπεζική ένωση που σχεδιάζει το συμβούλιο η επιτροπή η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και δυστυχώς η σημερινή πλειοψηφία του κοινοβουλίου δίνει συγχωροχάρτη στο τραπεζικό σύστημα που έχει τεράστια ευθύνη για την οικονομική κατάσταση στην ευρώπη σήμερα. αντί για ευκαιρίες ανάκαμψης και ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες η τραπεζική ένωση που σχεδιάζεται ενισχύει τις τράπεζες ζόμπι ενισχύει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα συνεχίσει να γεννά φούσκες ανισορροπία και κρίσεις. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Έλμαρ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η πρόταση που έχουμε σήμερα στα χέρια μας είναι τελείως άστοχες για την Ευρωζώνη και τελείως άστοχες και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χωρί σύστημα εγγύσεω των καταθέσεων για τι τράπεζε τη Ευρωζώνη και γενικότερα, δεν θα υπάρχει κανένα, κανένα αποτέλεσμα. Και βεβαίω οι Γερμανοί δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα, διότι δεν θέλουν να καταλήξουν να διασώζουν τι τράπεζε των υπόλοιπων τραπεζών. Ούτε εμεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλουμε το City του Λονδίνου να χάνει χρόνο και εργασίε λόγω του περίπλοκου συστήματο νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τόσα διαφορετικά συστήματα, αλληλοσυμψηφισμού, διασώσει με ιδέα μέσα και άλλα τέτοια μπερδεμένα συγκεκριμένα μέτρα, τελικά δημιουργούμε ένα καρκίνωμα που είναι η ίδια η Ευρωζώνη. Ένα αποτυχημένο εγχείρημα που δεν έχει, κάνει ποτέ, ε, κανένα, δεν έχει φέρει ποτέ κανένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτή η ισχυρογνωμοσύνη των Ευρωπαίων ηγετών που δεν μπορούν να ε, αποδεχτούν την κατάρρευση του ε, δικού του συστήματο και του εγχειρήματο του ευρώ οδηγεί σε απελπισία την νεολαία στον νότο τη Ευρώπη. Φτάνει, κυρία Πρόεδρε, πρέπει επιτέλου να δοθεί ένα τέρμα σε αυτή την ανοησία του ευρώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Χέλμερ. Υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Δέχεστε την ερώτηση. Με μεγάλη μου χαρά. Κύριε Χέλμερ, εάν πιστεύετε ότι αυτές οι προτάσεις είναι τόσο άστοχες και τόσο απαράδεκτες, γιατί τότε η ομάδα σας δεν προσήλθε σε καμία από τις εκατοντάδες ε, συνεδρίες ε, διαπραγματεύσεων που είχαμε την τελευταία πενταετία για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα Δηλαδή το αποτυχημένο τραπεζικό μας σύστημα να το ρυθμίσουμε σωστά. Και γιατί περιμένετε την ακροτελεύτια σύνοδο ολομέλειας αυτού του Ευρωκοινοβουλίου μέχρι επιτέλους να υψώσετε τη φωνή σας. Γιατί. Uh, σε ευχαριστώ, Βίκη. Είναι πάντοτε ευχάριστο να ακούει κανεί ε, τι δικέ σου σκέψει. Σε μια μικρή ομάδα κανεί και σε θέση μειονότητα, όταν είναι μια ομάδα ευρωσκεπτικιστών που αντιτίθεται στο όλο εγχείρημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να παρακολουθεί η ομάδα αυτή κατά λεπτό τι εξελίξει των διαπραγματεύσεων, όσο σημαντικέ κι αν είναι. Και ε, βεβαίω ε, ήταν πολύ καλή ευκαιρία στο και σήμερα να εκφραστούμε για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστώ, Βίκη, που έθιξε και αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκοζές για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, είναι μεγάλη μου χαρά που όπως και περισσότεροι εδώ σήμερα ε, παρά τις κάποιες ε, μικρές ε, παραφωνίες. Μπορώ να ενώσω τη φωνή μου με αυτούς που συνεχάρισαν τον Επίτροπο για τη δουλειά τους. Αλλά και από την πλευρά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η σωστή αυτή ε, συνεργασία οδήγησε σε ένα σύστημα που νομίζω θα είναι μεγάλη αποτελεσματικότητα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να χαιρετήσω τι προσπάθειε όλων όσων συνέβαλαν, ώστε τα κείμενα αυτά να είναι έτοιμα πριν το τέλο τη θητεία και ώστε να ε, σεβαστούμε και το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα σε ένα αρκετά ε, δυσχερέ οικονομικό πλαίσιο. Στη διάρκεια αυτή τη θητεία καταφέραμε να δημιουργήσουμε του πυλώνε τη Τραπεζική Ένωση και του μηχανικού εποπτεία των τραπεζών με ένα σύστημα εξυγίανση και ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανση και σύστημα αγγίσεω των καταθέσεων με πολύ καλό τρόπο. Όλα αυτά τα κείμενα τελικό στόχο έχουν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, την εμπιστοσύνη του στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και να του προστατεύσουμε από του κινδύνου των τραπεζικών τριγμών. Εδώ λοιπόν όχι μόνο η δουλειά του Κοινοβουλίου ήταν σημαντική για την χρηματοπιστωτική, χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά ολόκληρη προσπάθεια η οικονομία να προστατευτεί από μελλοντικέ συστημικέ κρίσει ε, και οι χρηματαγορέ και οι τράπεζε να αρχίσουν επιτέλου να υπηρετούν την πραγματική οικονομία. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τι διαφωνίε μα ε, με τη γενικότερη αντίληψή μα για την τραπεζική ε, για την Τραπεζική Ένωση ή για το ενοποιημένο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων αυτό αποδεικνύει τι συλλογικέ μα προσπάθειε να καταλήξουμε σε καλύτερε λύσει. Και τι λύσει αυτέ, επίτροπε, σε μεγάλο μέρο τι συμμεριστήκατε και το εκφράσατε και στη σημερινή συζήτηση. Πραγματικά νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση είναι το κερασάκι στην τούρτα, αν μπορώ να το πω έτσι, σε μια νομοθετική διαδικασία που ήταν υποδειγματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπερές για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει υπερβολική ανεργία με 26 εκατομμύρια ανέργους. Εκαιρό είναι να ασχοληθούμε και με τις υπερβολές του τραπεζικού τομέα που έφεραν σε τόσο δυσμενή κατάσταση τα δημοσιονομικά των χωρών μας. Καλό είναι λοιπόν να εγκρίνουμε αυτά τα μέτρα για τη λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης με τρεις πυλώνες. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω, δεν το συνηθίζω, τον συνάδελφο Χόκμαρτ, γιατί με την έκθεσή του προτείνει τη διαδικασία εκείνη όπου μία τράπεζα σε δυσκολία πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της. Ο στόχος είναι απλός. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, οι καταθέτες δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή για να διασώσουν μια τράπεζα σε δυσκολία και αυτό από 1η Ιανουαρίου 2016. Είναι οι μέτοχοι και οι πιστωτές που κατά πρώτον αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις απώλειες των τραπεζών. Με την έγκριση λοιπόν της ε, έκθεσης Σίμων επίσης έχουμε και προστασία των καταθέσεων υπάρχει αναρμόνιση. Σε περίπτωση αποτυχίας μιας τράπεζας, οι Ευρωπαίοι πολίτες σε 7 μέρες μπορούν να έχουν μέχρι 100.000 από τις καταθέσεις τους. Είναι μια υπόσχεση που γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, έχουμε και την έκθεση της συναδέρφου Ελίζα Φερέρα. Εδώ πραγματικά βρισκόμαστε στο σκληρό πυρήνα. Έγινε μεγάλη, δόθηκε μεγάλη μάχη όλους αυτούς τους μήνες και ευχαριστώ για τη στήριξη της πολιτικής μου ομάδας στη συζήτηση αυτή. Γιατί έτσι αποδείξαμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση η οποία επιτρέπει να ξεπερνάμε τις προσεγγίσεις των χωρών μελών και που επιτρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας μια πραγματική τραπεζική ένωση και που καταστρέφεται πια αυτή η σχέση ανάμεσα στις τράπεζες και τα δημοσιονομικά των χωρών μελών. Επιτέλους μπορούμε έτσι να δώσουμε νεόθυση στις επενδύσεις. Τους ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν σε αυτό και επιτέλους μπαίνουμε στα σημαντικά που απασχολούν τους πολίτες μας που είναι οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κλούτα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν υπογραμμίζω και τονίζω ότι πιστεύουμε ότι η Τραπεζική Ένωση είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν θέλουμε ένα νόμισμα ενιαίο, θέλουμε και σαφή ρύθμιση του τραπεζικού τομέα και, συντονισμού της οικονομικής, και συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Το είπαμε και στην αρχή της κρίσης αυτό. Κάποιες ε, κριτικές παρατηρήσεις τώρα. Ο στόχος της Τραπεζικής Ένωσης είναι η προστασία των φορολογουμένων. Ε, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί η προοικοδότηση αυτού του μέσου δεν ξέρουμε αν θα είναι επαρκής. Θα το δούμε. Όμως έχουμε πολλές αμφιβολίες. Ίσως θα πρέπει να εργαστούμε στο μέλλον πάνω σε αυτό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μας είναι το πρόβλημα των too big to fail που δεν λύνεται ε, όπως το επιχειρούμε δεν είναι δυνατόν. Παραμένει μεγάλη πρόκληση το ζήτημα αυτό για την επόμενη θητεία των πολύ μεγάλων για να αποτύχουν. Ελπίζω να λύσουμε ικανοποιητικά το θέμα αυτό στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από πέντε χρόνια θητείας μπορούμε με μεγάλη περηφάνεια να πούμε ότι αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί το 2009 στους πολίτες, δηλαδή να δημιουργήσουμε σταθερές χρηματοοικονομικές αγορές, και να ελαφρύνουμε τον φορολογούμενο ε, προκειμένου περικρίσεων, αυτό το καθήκον το αντιμετωπίσαμε καλά. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκούς εποπτικούς μηχανισμούς, καταφέραμε στη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών, θα ψηφίσουμε απόψε, να ε, προβούμε σε πολλές ρυθμίσεις ούτως ώστε να μην έχουμε μη ρυθμιζόμενες αγορές και προϊόντα στα κράτη-μέλη. Τώρα με την Τραπεζική Ένωση ε, συμβάλλουμε ώστε ο ίδιος ο τομέας να αναλαμβάνει τους κινδύνους του και όχι ο φορολογούμενος, ο οποίος θα αποτελεί την ε, καταφυγή πρώτης γραμμής. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτό που καταφέραμε στα πλαίσια αυτής της θητείας του Κοινοβουλίου. Τώρα, για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα πω δύο λόγια, γιατί δυστυχώς στην ψηφοφορία δεν προβλέπεται απόψε συζήτηση. Ε, δυόμιση χρόνια συμμετείχα σε πολλές διαπραγματεύσεις, με πολλές προεδρίες, σε μακρές συνεδριάσεις με τον Επίτροπο. Ε, έπρεπε να ε, επεξεργαστούμε μια υποδειγματική λύση η οποία θα μπορούσε να ισχύει και σε άλλες χρηματοπιστωτικές αγορών εκτός Ευρώπης. Ευχαριστώ για την συνεργασία αυτή και τη συναδελφικότητα καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δωμένης, για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Αντζελίλη. Αυτή είναι η τελευταία σύνοδος ε, της θητείας μας στο Στρασβούργο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε και ένα γενικό απολογισμό για την ε, νομοθέτηση του τραπεζικού και οικονομικού τομέα που, που προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ νομίζω πως μπορούμε να πούμε και ναι και όχι. Διότι φωτίστηκε με πολύ καλό τρόπο στη συζήτηση το τι λύσεις προσπαθήσαμε να δώσουμε σε κάποια θέματα, αλλά υπήρξαν και κάποιες σκίες. Είναι θετικό απολογισμό τη εργασία των ε, εισηγητριών και εισηγητών για το μηχανισμό εξυγίανσης, το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, τη γενικότερη προσπάθεια που έγινε να προασπιστούμε τους πολίτες και του φορολογουμένους. Όμως δυστυχώς κάποιε φορέ οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα μακρο, μακρές για να ε, ε, υλοποιήσουμε τους κανόνες που προβλέπουμε και λυπούμε που σε αυτή τη θητεία δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και το εγχείρημα του διαχωρισμού των ε, επενδυτικών τραπεζών και των εμπορικών. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας από τους πρώτους στόχους της ευερχόμενης θητείας. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο την ε, τάση των τραπεζών ε, να διωγγώνουν την προσφορά τους και των υπηρεσιών τους. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικότερη διαχείριση στις τράπεζες ώστε να ελέγχουμε τι κάνουν τα ανώτατα στελέχη των τραπεζών και ιδίω με τι τράπεζε τι συνεργατικέ που δρούν στην πράξη και όταν η συνεργασία ξεπερνά τα σύνορα ενό κράτου μέλου. Θα πρέπει να εγγυθούμε την σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματο ε, σε ένα εθνικό σύστημα. Όπω έλεγε και ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, είναι καλύτερη πρόληψη παρά η θεραπεία όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόεδρος, η κυρία Ποδηματά για 1,5 λεπτό. Πολύ, κυρία Πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό και έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό ότι σε αυτήν την τελευταία μας ολομέλεια επικυρώνουμε τη συμφωνία για το δεύτερο πυλώνα της τραπεζικής ένωσης τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών ε, μαζί με το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης που μαζί με τον ε, ενιαίο εποπτικό μηχανισμό θέτουν τις βάσεις για την άρση του κατακαιρματισμού και των επικίνδυνων ανισορροπιών του τραπεζικού συστήματος της ευρώπης και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υγιείς τράπεζες με ενιαίους και διαφανείς κανόνες εποπτείας λειτουργίας και εξυγίανσης όταν και εφόσον χρειαστεί σημαίνει όχι μόνο προστασία των φορολογουμένων από βάρη που δεν τους αναλογούν σημαίνει και ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της ρευστότητας και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και χαίρομαι για τη μεγάλη συμβολή της ελληνικής προεδρίας στην επίτευξη συμφωνίας και χαίρομαι ιδιαιτέρως κύριε προεδρεύοντα του συμβουλίου που υπενθυμίσατε πολύ σωστά ότι η τραπεζική ένωση έχει και έναν τρίτο πυλώνα που δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ε, η δρομολόγηση του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων με ένα ενιαίο ταμείο στα πρότυπα του ενιαίου ταμείου ε, εκαθάρισης ελπίζω επίτροπε μπαρνιέ και σας ευχαριστώ με την ευκαιρία για το εξαιρετικό έργο σας συνολικά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην τραπεζική ένωση ότι η επόμενη ευρωπαϊκή επιτροπή θα δεσμευτεί να προχωρήσει και να υλοποιήσει και αυτόν τον τρίτο απολύτως απαραίτητο πυλώνα της τραπεζικής ένωσης. σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τάισεν έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από την αρχή της θητείας αυτής δεν φανταζόμασταν ότι θα καταφέρναμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο με τον ενίο εποπτικό μηχανισμό, με τον μηχανισμό εκαθάρισης και με το σύστημα για τις εγγύησεις καταθέσεων. Τα καταφέραμε και πρέπει να είμαστε περήφανοι για το έργο μας. Οι προσπάθειές μας για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω ενός φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού σχεδίου βοήθησαν την Ευρώπη να πάει μπροστά. Η συνεργασία μας στο σώμα αυτό, αλλά και συνεργασία με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους ιδιαίτερος με την ομάδα του κύριου Μπαρνιέ οδήγησε σε αποτελέσματα και το θαύμα έγινε πραγματικότητα. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε περήφανοι. Περήφανοι για τις επιτυχίες μας όσον αφορά τα αντανακλαστικά των χωρών, για τους μηχανισμούς που πετύχαμε, για τον ενίο μηχανισμό που αντιμετωπίζει τις τράπεζες και για χώρες εκτός της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ασφαλές οικονομικό σύστημα που να μπορεί να προχωρήσει σε καθάριση των τραπεζών, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα, εξασφαλίζοντας κανόνες που να βοηθούν όλους τους πολίτες. Αυτά τα νέα μέτρα λοιπόν τώρα έρχονται στα πλαίσια μια νέας προοπτικής, πια ξέρουμε τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες και τι ρόλο πρέπει να παίζουν στην πραγματική οικονομία που είναι να προσφέρουν ρευστότητα και θέσεις απασχόλησης. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλους. Χάρη στη συνεργασία αυτή φτάνουμε στα σημερινά αποτελέσματα και τέτοια συνεργασία χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να είμαστε σχηροί ισχυρή ανάμεσα στον κόσμο ολόκληρο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καράς για δύο λεπτά τώρα. Κύριε Πίτροπε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα καταφέραμε και τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Σήμερα ένα πρόγραμμα μαμούθ ε, αποφασίζεται για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Έγινε το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση και δίνονται διασφαλίσεις για τους πολίτες της Ένωσης. Η Τραπεζική Ένωση ε, σημαίνει ότι σε περίπτωση πτωχεύσεων δεν θα βάζουμε χέρι στην τσέπη των φορολογουμένων και καταθετών. Έτσι κάνουμε σταθερότερη την Ένωση και πιο ανθεκτική στις κρίσεις. Η νέα ρύθμιση ιδίων κεφαλαίων δημιουργεί πρότυπα και κανόνες για όλες τις τράπεζες. Η κοινή εποπτεία της ε, ΕΚΤ ε, σημαίνει ότι θα υπάρχουν ίσοι όροι ε, για όλους. Υπάρχει το δίκαιο πτωχεύσεων τραπεζών που ρυθμίζει τις διαδικασίες για όλες τις τράπεζες. Προβλέπεται ταχεία εκταμίευση των καταθέσεων των μικροκαταθετών. Ε, εκεί στηρίζεται το ε, Ταμείο Προστασίας Καταθετών. Το Μπέιλιν, διάσωση με ίδια μέσα, ε, θα στηρίζεται και στο δημιουργούμενο Ταμείο Εκαθάρισης. Δεν θα χρησιμοποιούνται πια τα χρήματα των φορολογουμένων για τη διάσωση ε, πτωχευμένων τραπεζών. Στη Βασιλεία 3 ε, έχουμε και αποφασίσει και ε, εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν επίσης λεπτομερή κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται. Εμείς ως νομοθέτες έχουμε δημιουργήσει σαφείς κανόνες και θέλουμε οι αποπτικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη συνεπή εφαρμογή των νέων διατάξεων. Ε, αν θεωρεί μια τράπεζα ε, ότι ε, δεν διατρέχει κίνδυνο στα πλαίσια του κανονισμού θα πρέπει να, να το κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές. Ε, εδώ υπάρχει στην πρότασή σας ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν θέλουμε να μείνουν κενά, δεν θα τα ανεχθούμε τα κενά. Θέλουμε να ε, εφαρμοστεί η, ε, ο να, εφαρμοστούν οι κανόνες για τις τράπεζες 100% για να εξαλειφθούν όλα τα κενά και τα ερωτηματικά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στόλογιαν για μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ όλες τις εισηγήτριες και τους εισηγητές που εργάστηκαν για αυτό το τόσο σημαντικό νομοθέτημα, ώστε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση της Τραπεζική Ένωση. Θέλω όμω να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω τον Επίτροπο Μπαρνιέ, για τι άκοπε προσπάθειέ του να καταφέρουμε να πείσουμε όλοι μαζί όσους δεν πιστεύουν στην δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύνει προβλήματα. Να τους θυμίσω την αλήθεια αυτή που εμπεριέχεται στη δήλωση του Σούμαν ε, στην στιγμή που ιδρυόταν η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η Ενωμένη Ευρώπη είναι κάτι που δεν το πετύχουμε εν μία νυχτή και με μία και μόνο λύση διαδικασία, αλλά με μικρά σταθερά βήματα που θα δημιουργήσουν μία de facto αλληλεγγύη. Πιστεύω ότι η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία με την πρόταση του ΕΛΚ να αλλάξει η συνθήκη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά απεικονίζει όλη αυτή την πρόοδο που έχουμε επιτελέσει προς την δημιουργία μιας πραγματικής νομισματικής, τραπεζικής αλλά και οικονομικής ένωσης. Πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να οδηγηθούμε σε ακόμη μεγαλύτερη σύγκληση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Φέγιου για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, σήμερα σε αυτή τη συνοβολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ζούμε μια ημέρα ιστορική. Η συζήτηση για το θέμα της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι ιστορική, αλλά το ίδιο και η ψηφοφορία όλων αυτών των νομοθετικών κειμένων που είναι ουσιαστικής σημασίας. Γι' αυτό θέλω πραγματικά να συγχαρώ το Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω τον Επιτροπό Μπαρνιέ, αλλά και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μπαρόζο και το Συμβούλιο για όλες τις προσπάθειες που έγιναν για το θέμα αυτό. Μια από τις υποσχέσεις που πολλοί από εμάς αναλάβαμε το 2009 είναι ότι δεν θα πρέπει πλέον οι φορολογούμενοι να πληρώνουν, να πληρώνουν για προβλήματα τραπεζικής φύσης. Σήμερα επιτέλους αποστέλουμε ένα σαφέστατο μήνυμα ως προς αυτό το θέμα. Τη σελίδα αυτή την έχουμε πλέον γυρίσει. Η Τραπεζική Ένωση είναι μια θετική ευρωπαϊκή απόκριση. Επιπλέον, ε, η τόκοι που θα πρέπει να πληρώνουν οι επιχειρήσεις για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν θα πρέπει επιτέλους να εξισώνονται γιατί θα πρέπει ακριβώς αυτά που ε, αναλαμβάνονται ως κίνδυνος να καταβάλλονται από τους υπεύθυνους, όχι οι καταθέτες να πληρώνουν τη λυπητερή. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και η νέα θητεία μετά τις ευρωεκλογές. Και αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση ως Ευρωβουλευτού. Θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ από καρδιά τα πάντα να πάνε καλά στην επόμενη θητεία, ώστε να συνεχιστεί αυτή η θετική κατεύθυνση στην προσπάθεια προστασία των καταθετών. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή για όλα όσα έκαναν για την Ευρώπη, για όλη τη στήριξη που έδωσαν σε αυτή τη διάρκεια τη θητεία και για όλη την πολιτική ανάπτυξη που πετύχαμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Πραγματικά ελπίζω αυτή η προσπάθεια και αυτή η κατεύθυνση να συνεχιστούν αμύωτες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο. ευχαριστούμε κυρία Χίμπνερ για 1,5 λεπτό. Uh, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ όλους όσοι έλαβαν ε, μέρος στις διεργασίες για να καταλήξουμε στα νομοθετήματα αυτά για την Τραπεζική Ένωση. Και ευχαριστώ πολύ που διατηρείται η ενιαία αγορά και δεν βαθύνονται περισσότερα τα χάσματα. Οι φορολογούμενοι λοιπόν προστατεύονται τώρα όταν οι τράπεζες αποτυχαίνουν. Το ενιαίο ταμείο θα βοηθάει να δανείζεται στην κεφαλαϊκή αγορά και να αντισταθμίζει έτσι το γεγονός ότι οι χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη δεν έχουν πρόσβαση στο ECM. Τώρα πετυχαίνουμε καλή μεταχείριση και όσων βρίσκονται εκτός του συστήματος. Το σύστημα αυτό με το ενιαίο ταμείο είναι κάτι θετικό, γιατί έτσι ισχυροποιείται η δημοκρατική νομιμότητα. Και ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγένση. Είναι θετικό το ότι καταφέραμε να δώσουμε νέα ισορροπία. Και η οδηγία αυτή και οι εγγύσεις καταθέσεων θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα και τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ευχαριστούμε, Λάγγεν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά για το έργο του της περασμένης πενταετίας. Θυμάμαι πολύ καλά ότι ο προκάτοχός του, ο κύριος Μακρύβη, στις 15 Μαρτίου του 2009 είχε υποβάλει τις πρώτες προτάσεις γιατί ε, είχε πάει προηγουμένως στις υποδρομίες στην Ιρλανδία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μπαρνιέ. Η Τραπεζική Ένωση βέβαια δεν πρόκειται να αποβεί πανάκια, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά το Ταμείο Εκαθάρισης, ε, εδώ ε, η νομική βάση ήταν διαφορετική από αυτή που ζήτησε η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Γιατί το Ταμείο Εκαθάρισης Τραπεζών δεν θα λύσει ε, τις παλιές περιπτώσεις, μόνο τις μελλοντικέ. Οι άλλες θα ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε πρόκειται για την τέξη στο Μπενελούξ, είτε στη Γερμανία την ΑΕΗ ή την Κρεντή Αγκρικόλ στη Γαλλία. Το Ταμείο Εκαθάρισης δεν θα τις λύσει αυτές, η πρικοδότηση με ίδια κεφάλαια κλπ. Όμως χαίρομαι διότι οι καταθέσεις αντιμετωπίζονται με νέο τρόπο. Όμως δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Ταμείο που θα καλύπτει τις καταθέσεις. Ε, όταν ε, υπάρχουν ε, εύρωστες καταθέσεις σε ένα κράτος μέλος δεν θα υπάρχει ευθύνη για προβληματικές τράπεζες αλλού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τέλος επέμεινε τα stress πριν από την ανάληψη της ευθύνης να γίνονται πάντοτε. Γι' αυτό είναι σημαντική η Τραπεζική Ένωση, αλλά όπως είπα δεν αποτελεί πανάκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα διαδικασία καθιάει. Δέκα είναι οι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο. Απλώς θα πρέπει να σεβαστείτε το μονόλεπτο χρόνο ομιλίας. Μαγκίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Γκούναρ, Μαριάννη, Κορίν, και όλοι οι υπόλοιποι, σε όλε τι πολιτικέ ομάδε, για αυτή την εξαιρετική δουλειά που συζητούμε σήμερα. Επίτροπε, είπατε ότι η κρίση αυτή ήταν οξία οξία ήταν πραγματικά ως προς τις επιπτώσεις που είχε στις οικογένειες, στην κοινωνία, στην πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε τους αριθμούς, αλλά να θυμίσω απλώς τι συμβαίνει στην Ιρλανδία. Στη δική μας τη χώρα οι φορολογούμενοι δέχτηκαν το πλήγμα και είπαμε αυτό να μην ξανασυμβεί ποτέ στο μέλλον. 64 δις ευρώ ήταν το κόστος. Εδώ χαιρετίζουμε τη συμφωνία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από τον Ιούνιο του 2011 ώστε να διαρριχθεί ο δεσμός μεταξύ κρατικού χρέους και τραπεζικών χρεών. Και αυτή η υπόσχεση πραγματικά ε, εκπληρώθηκε ως προς την Ιρλανδία. Ευχαριστώ λοιπόν για το ήθος σας Επίτροπε και για την ευθύνη σας. Δεν είναι η πρώτη φορά και σας ευχαριστώ που χρησιμοποίησατε αυτά τα λόγια στην αίθουσα της Ολομέλειας για τον τραπεζικό τομέα. Καλή τύχη λοιπόν σε όσους θα εκλεγούν στο μέλλον και σε όσους δεν θα ξαναδούμε εδώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλλη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπαν όλοι, είναι μια σημαντικότατη ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. φτάνουμε στο τέλος μιας πενταετίας δουλειάς, σκληρής δουλειάς. Και θέλω να επενέσω όλους τους συναδελφούς, αλλά και τον Επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ, διότι Νομίζω ότι πραγματικά θα μπορέσετε να αναλάβετε ένα αξίωμα που να αρμόζει και στι ικανότητέ σα, όπω το αποδείξατε την τελευταία πενταετία. Ήθελα εδώ να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, το σύστημα εγγύηση καταθέσεων είναι ένα τεράστιο σύστημα. Πολύ σημαντικό για του καταθέτε για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη προ τι τράπεζε. Πολύ καλή η δουλειά που έγινε εδώ. Εδώ, επίση, οι ε, δυνατότητε ε, συνεργασία των τραπεζών έχουν περιοριστεί, ώστε τα πράγματα να είναι τουλάχιστον λίγο πιο ρυθμισμένα από ό,τι στο μέλλον. Και επίση, ο φόβο ότι μπορεί να είναι πολύ μεγάλη τραπεζική όμιλη αναφέρθηκε. Ναι, δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλε οι τράπεζε ώστε να μην αποτυγχάνουν. Στην Ιρλανδική περίπτωση αυτό επιβεβαιώθηκε και γι' αυτό θέλω να σα ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε. Πλάνκοβιτ. Πρόεδρε, χαιρετίζω την παρουσία του κύριου Μπαρνιέ και εκφράζω το σεβασμό μου για την δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια ολόκληρη της κρίσης αυτής. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους δύο εισηγητές με τις δύο προτάσεις τους που επιτρέπουν να συμπληρώσουμε έτσι την Τραπεζική Ένωση και να στείλουμε το μήνυμα που λέει ότι τελικά η Ευρώπη κάνει αυτό που πρέπει και δεν ισχύει το ότι ό,τι κάνει το κάνει πολύ αργά. Έτσι έχουμε μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα. Και ελαχιστοποιούμε επίσης και το κόστος που επομίζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες σε περίπτωση αποτυχίας τραπεζών που είναι αφαιρέγγες. Πιστεύω ότι με τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται θα ενισχύσουμε το επίπεδο προστασίας των πολιτών, αλλά και την εμπιστοσύνη τους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πρέντεργκαστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θέλω να αποτίσω φορό τιμή στην δουλειά που έγινε από την κυρία Φερέρα, στην ε, πραγματικά αφουσιωσή τη και την επιμονή τη παρά τι επανελειμμένε αποτυχίε του οικονομικού τομέα να κάνει τόση δουλειά από το 2008. Όπω είπαν τόσοι συνάδελφοι, μα κόστησε 64 δι ε, δημοσίου χρήματο, δηλαδή τέσσερι κοινοτικού προπολογισμού. Την ημέρα αυτή πετυχαίνουμε ένα βήμα προόδου για μια ισχυρότερη και πιο συνετή τραπεζική διαχείριση. Δηλαδή δηλαδή να έχουμε καλύτερη εποπτεία για τις ε, τράπεζες και περισσότερες απαιτήσει για τα κεφάλαια. Τουλάχιστον παίρνουμε τη σωστή κατεύθυνση για την αναδιάρθρωση των ε, τραπεζών μας. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο νομοθέτημα που θα έχει περάσει από αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία. Πραγματικά εύχομαι να τα έχουμε καταφέρει να το ολοκληρώσουμε νωρίτερα και τα κράτη-μέλη να πάνε ακόμη παραπέρα. Υπάρχει σωστή ιεράρχηση των μετόχων και των ομολογιούχων που δεν θα ε, επιβάλλουν πλέον στους φορολογουμένους τις απώλειες των τραπεζών. Επιτέλους θα μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μάνκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2006 οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είχαν υποβάλει ήδη προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων. Όμως οι ευρωσκεπτικιστές και το Ευρωκοινοβούλιο τότε είχαν απορρίψει τις προτάσεις αυτές λέγοντας ότι θα αυτορυθμιστεί εφόσον χρειαστεί η αγορά. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε ότι χρειάστηκε τις τράπεζες να τις σώσουν αυτοί που δεν ήταν υπεύθυνοι για τα προβλήματά τους. Θα ήταν ωραία αν όλα ήταν ιδανικά στην αγορά και τα κέρδη κατανέμονταν ε, ισότιμα μεταξύ των ε, ε, όσων θα έπρεπε να λάβουν όφελο. Όμω δεν συμβαίνει αυτό. Το κέρδο το παίρνουν λίγοι και τι ζημιέ τι πληρώνουν ε, αυτοί που δεν φταίνε. Τώρα το σύστημα γύση των καταθέσεων ε, δείχνει ότι δεν θα πληρώνουν πλέον οι φορολογούμενοι, αν και κανεί δεν του προστατεύει ε, πλήρω από τι ζημιέ. Ούτε οι οι τραπεζίτε ούτε οι μέτοχοι μπορεί να είναι προστατευμένοι από τον κίνδυνο αποτυχία. Θα πρέπει να ελέγχουν και να διαχειρίζονται καλύτερα τι τραπεζέ του. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα διανύουμε στην Κύπρο την εβδομάδα των παθών, προσδοκώντας το Πάσχα και την Ανάσταση. Την ίδια ώρα, εδώ στο Στρασβούργο, κάνουμε ένα απολογισμό πενταετίας για όσα πράξαμε ή παραλείψαμε για να αντιμετωπίσουμε τα κενά και τις αδυναμίες που ανέδειξε η οικονομική κρίση. δυστυχώς ο απολογισμός είναι θλιβερός γιατί εμείς οι κύπροι πολίτες γίναμε τα πειραματόζωα για να δούμε σήμερα πώς αντιμετωπίζουμε το συστημικό κίνδυνο πώς η ανυπαρξία κανόνων και μέσων γίνεται σήμερα νομοθεσία πώς αντιμετωπίζεται η χρεοκοπία τραπεζών δυστυχώς βλέπουμε σήμερα πως γίνεται μια προσπάθεια για το μέλλον. τι γίνεται όμως για τη δική μου πατρίδα την κύπρο για τους πολίτες της που βιώνουν ακριβώς όχι μόνο αυτή τη βδομάδα τα πάθη αλλά του, τελευταίους μήνες. πότε θα έρθει η ανάσταση αφού αυτά που σκεφτόμαστε είναι για το μέλλον δεν είναι για το χτες και τα λάθη που έκαναν οι ευρωπαίοι. Ευχαριστούμε, Ευχαριστώ. Η σταθερότητα του ευρωπαϊκού τομέα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να έρχεται πριν από την προστασία των φορολογούμενων. Γιατί ανεύθυνες κυβερνήτες συζήτησαν τη δικιά τους βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την κρίση για το δημόσιο χρέος. Μια τέτοια πολιτική βόλευε τις τράπεζες γιατί δημιουργούσε νέα χρέη και έτσι στήριζε την αποτυχημένη αυτή πολιτική. Έτσι οι τράπεζες συμμετείχαν στην αναδιάρθρωση. Σήμερα θέλουμε να προστατεύσουμε βέβαια τις αποτυχημένες τράπεζες, αλλά πρώτα απ' όλα τους φορολογούμενους και τους μικροκαταθέτες από μια αποτυχημένη πολιτική η οποία χρηματοδοτείται με δικά τους χρήματα. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που διαπιστώνω ότι σύμφωνα με την πρόταση αυτή οι πόροι για τη διάσωση των τραπεζών δεν προέρχονται από τους προπολογισμού των χωρών μελών και γι' αυτό και την υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Βούλγανιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν είναι ιστορική σημασία σήμερα αυτή που λέμε ότι πρέπει να πληρώνουν αυτοί που δημιούργησαν την κρίση. Όχι, η κρίση είναι αποτέλεσμα μιας ανεύθυνης συμπεριφοράς τράπεζας και της πολιτικής τους της πιστοτικής, όπου οι τράπεζες χρησιμοποιούν χρήμα που δεν διαθέτουν στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εφ' θα αλλάξουν τα πράγματα, δεν θα πληρώνει ο φορολογούμενος. Όμως ο κίνδυνος παραμένει ο τραπεζικός τομέας να παραμένει κράτος αν κράτη, που διαχειρίζεται τα χρήματά μας για να δημιουργήσει εικονικό χρήμα, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δηλαδή. Ελπίζουμε ότι η επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να δουλεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Λαβράκοφ. Είναι θετικό να υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μήνυμο εγγύσεων της αποταμίευσης της μικράς και μεσαίας τάξης καταδετών και η αύξηση των προσβλέψεων των τραπεζών για επισφαλείς απαιτήσει. θεωρώ επιτυχή την προσπάθεια παρότι φοβάμαι ότι το θέμα της οικονομικής κρίσης μεταφέρεται και πάλι στους φορολογούμενους πολίτες πολίτες καταθέτες και όχι στους μετόχους αλλά κυρίως μακράν της εποπτείας που έχει τις ευθύνες της. πέντε χρόνια τώρα υποκρινόμεθα ότι αγνοούμε ότι η κρίση είναι και νομισματική η κεντρική μας τράπεζα πρέπει να λάβει επιπλέον μέτρα νομισματικής χαλάρωσης για να αντιμετωπιστεί ο χαμηλός πληθωρισμός και το ισχυρό ευρώ που βάζουν φρένο στην ανάπτυξη της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα της πλειοψηφίας των κρατών μελών. θεωρώ ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αντιστοιχία του ευρώ με το δολάριο που ανατράπηκε μετά την έκδοση των έξι τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τη σύπα με την ευκαιρία ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και κυρίως και τον επίτροπο μπαρνιέ για την προσπάθεια την οποία έχει κάνει στα θέματα του χαρτοφυλακίου του και τη συνεργασία που είχαμε. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μοργάντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε λέγεται ότι σε περιπτώσει κρίση έχουμε υποχρέωση να σώσουμε τι τράπεζε γιατί τελειώς να καταρρεύσει όλο το οικονομικό σύστημα. Αληθεύει αυτό. Αλλά μόνο και μόνο γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο χωρί επιστροφή όπου οι τράπεζε γίναν τερά... τεράστιου όγκου και η πτώχευσή του θα μπορούσε να... να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Χρησιμοποιήσαμε κατά τρόπο μαζικό τι αποταμιεύσει των ε, καταθετών μέχρι τώρα, των απλών πολιτών και θα πρέπει επιτέλου να προστατεύσουμε του καταθέτε, του απλού φορολογούμενου. Δεν είχαμε την τόλμη να αναλάβουμε μέτρα πριν όλα αυτά συμβούν. Ε, Επίτροπε Μπαρνιέ, αναφέρομαι στον σαφή διαχωρισμό των ε, τραπεζών βάσει του μοντέλου τη Αμερική από το 1933. Η ιστορία θα πρέπει κάτι να μα διδάξει. Ότι δηλαδή είχαμε ένα παράδειγμα για το τι θα πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από αυτήν την κρίση. Οι τράπεζε πρέπει να παραμείνουν τράπεζε. Δηλαδή να δέχονται αποταμιεύσει και να διαχειρίζονται τι οικονομίε των πολιτών πολιτών για να λειτουργεί πραγματική οικονομία. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θέλουν να αναλαμβάνουν κίνδυνο και να κερδοσκοπούν στι αγορέ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Μπορούν να το κάνουν, αλλά όχι με τα δικά μα χρήματα ή με τι δικέ μα εγγυήσει. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διανύσαμε ένα μακρύ δρόμο μαζί. Ήμασταν 28. Το λέω αυτό για την προηγούμενη παρατήρηση για το City του Λονδίνου. Δεν είναι τυχαίο που ήμασταν 28. Ήταν ε, εθελοντική η δουλειά που έγινε, όγκο τη δουλειά που έγινε από τη δική μου την πλευρά, αλλά και από τι δικέ σα τι κυβερνήσει, για να στηρίξουμε την εσωτερική αγορά και βεβαίως και με αυτή την τεράστια χρηματαγορά, αυτό το city του Λονδίνου, το οποίο σεβόμαστε όλοι. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι βουλευτές, το λέω, διότι κάποιοι είπαν ότι ήρθαμε πολύ αργά στην Τραπεζική Ένωση. Χρειάστηκαν διαφορετικέ μεταρρυθμίσει εδώ και θυμίζω ότι η δική μου προτεραιότητα, όλων μα προτεραιότητα, ήταν να δημιουργηθούν τρει αρχέ εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, την, ε, με όλη τη συνεργασία όλων ε, των Ευρωβουλευτών Γκουλάρ, Σκίνερ, ε, Μαριέλο και ούτω καθεξής καταφέραμε πολύ γρήγορα μέσα σε δύο χρόνια για την Ευρωζώνη να καταφέρουμε αυτό που θέλαμε και όσοι θέλουν να έρθουν στην Τραπεζική Ένωση κάτι να καλώς να ορίσουν και η Σουηδία και ποια άλλη χώρα θέλει διότι είναι σαφές ότι η σταθεροποίηση της Ευρωζώνης ή η αστάθειά της, όπως είδαμε τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι σταθερότητα, σταθερότητα ή αστάθειας ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η Τραπεζική Ένωση είναι πραγματικά ουσιαστικής σημασίας. Η κυρία Φερέιρα, η κυρία Τάισεν και ο κύριο Γκίγκολτ εργάστηκαν πολύ σκληρά για αυτά τα θέματα, αλλά όπω είπε και η κυρία Βορτμαν Κόλ, θέλω να χαιρετήσω και τον ιδιαίτερο ρόλο τη Ελληνική Προεδρία ε, και του προέδρου του ε, Eurogroup, του κύριου Δίσεμπλουμ, και βεβαίω τον κεντρικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Ακριβώ Τράπεζα σε όλε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Με την ε, αντιπροεδρία του Βίκτορ Κοντάντσιου. Και να πω ότι έχουμε πλέον κοινού κανόνες ώστε να γλιτώσουμε τους καταναλωτές, τους πολίτες. Δεν θα πληρώνουν πλέον ε, για τι τράπεζε με την οδηγία BRD, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένω ο συνάδελφο Και με κανόνες προληπτικούς, διαρθρωτικού, ώστε όλοι οι παράγοντε της αγοράς το είπε ο κύριος Μπάλς προηγουμένως, αλλά και ο κύριος Κάρας, ε, είναι σημαντικά αυτά και διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο για τις 3.500 τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για διορθωτικέ αλλαγέ για να περιορίσουμε τους κινδύνους, για να υπάρχει μια ε, σωστή εποπτεία, για να υπάρχει ανάληψη ευθύνη. Και πρώτη κλίδα για την ανάληψη ευθύνη είναι η διαφάνεια, δηλαδή ποιο κάνει τι. Εμείς φωτίσαμε, φωτίσαμε αυτές τις πτυχές για ανθρώπους που δεν τα βλέπουν τόσο ξεκάθαρα και πρέπει να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε, γιατί Μαρέιτ Μαγκίνε, μίλησε για ήθο και για διοντολογία πολύ σωστά αναφέρθηκες και σε, αυτά, σε αυτές τις έννοιες. Διότι πρέπει να μιλάμε για τέτοιες έννοιες όταν νομοθετούμε και μιλάμε για θεμελιώδεις νομοθετικές πράξεις. Και όταν μιλάμε στους πολίτες για ήθος και δεντολογία αλλά και για κίνδυνο και γι' αυτό απαντώ εδώ στον ε, κύριο Κάρας για τη συγκεκριμένη παρατηρήση που έκανε για τους τεχνικούς κανόνες των αμοιβών Είναι σημαντικό και αυτό. Να χαιρετήσω εδώ την προσπάθειά σας πριν από λίγες εβδομάδες για τους τεχνικούς κανόνες για τις αμοιβέ που ισχύουν στην περίπτωση ε, των ειδικών ε, συνεργατών. Και επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις προσπάθειες που έκαναν. Ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο. Και όντως οι αρχές του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει εξάντε να ε, ενημερώνονται για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και για την ερμηνεία των τεχνικών κανόνων και για τη δική σας ερμηνεία κύριε Κάρας με την επίσημη επιστολή σας. Είναι ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα όπου ανέμεναν απαντήσεις οι πολίτες και εσείς ως βουλευτές τις δώσατε. Τις δώσατε βάσει του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της συνεργασίας του Συμβουλίου. Διότι δεν μπορεί ο κόσμος της οικονομίας να θεωρεί ότι όλα το επιτρέπονται, ούτε να τους τα επιτρέπουμε όλα όπως συνέβαινε πριν από 25-30 χρόνια. Θα πρέπει ο κόσμος οικονομία, όπω ο κύριο Γκοζέ, να εξυπηρετεί πλέον την πραγματική οικονομία, όχι τον εαυτό του. Εργαστήκαμε σκληρά. Και επειδή μιλώ για τους πολίτες και τους φορολογουμένους, αυτούς θελήσαμε να προστατεύσουμε. Και εδώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να θυμίσω κάποια νομοθετήματα που υιοθετήσαμε πριν από εδώ και τέσσερα χρόνια. Κείμενα για τους πολίτες. Η εγγύηση των καταθέσεων. Είναι για τους πολίτες κύριε Σίμων. Τρίψ, κύριε Μπερές. Ο βασικός τραπεζικός λογαριασμός, κύριε Κλούτα. Και ε, χαιρετώ εδώ και τη συνεργάτη δάμου που ήρθε και παρακολούθησε την εξέλιξη αυτής της, ε, ε αυτού του νομοθετήματος. τα ενυπόθηκα δάνεια, η, η πρόταση του κυρίου Σμιτ οι προτάσεις του κυρίου Φέγιο και Θάλμπα είναι κείμενα για τους πολίτες. Είναι κείμενα που επιτέλους αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν υποφέρει λόγω της κερδοσκοπίας και της εκμετάλλευσης είναι ε, καθοριστικά. Και εδώ πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η προσπάθεια για, αυτό το, ε, για αυτές τις ε, επιδιώξεις πρέπει να συνεχιστεί και για το private equity, οι προσπάθειες του κυρίου Γκοζές ήταν καθοριστικές, ε, αλλά και οι προτάσεις του κυρίου Αλκαντράουι. Για τα παράγωγα επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά σας. Εδώ μιλάμε για τομείς που σε όλο τον κόσμο 600.000 δις ευρώ είναι η αξία όλων αυτών των συναλλαγών στις διεθνείς χρηματαγορές. Πρέπει λοιπόν οι προσπάθειές μας να ε, συνεχιστούν αμύωτες. Οι προσπάθειες του κυρίου Λάμπερτς, οι καταχρήσεις στην αγορά, ε, ορισμένοι τραπεζίτες θα πάνε και φυλακή εφόσον υπάρχουν καταχρήσεις χάρη στην ε, πρόταση Μακάρθη και για τους οίκους αξιολόγηση με τον κύριο Ντομενίτσι, το Γιούσιτς με τον κύριο Γκίγκολ, ε, η πρόταση του κυρίου Καρίμ, η, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, οι προσπάθεια του κυρίου Λένε, η χρηματοοικονομική όμιλη του κυρίου Στόλογιαν και τόσα άλλα κείμενα που είναι σημαντικά για μένα και για την εσωτερική αγορά κείμενα που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη. Είναι το, διαβατά, το διαβατήριό όμω για τα κεφάλαια κινδύνου. Κύριε Λάμπερτ, κυρία Χιούμπνερ, τα αναλάβατε εσεί αυτά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τι κοινωνικέ επιχειρήσει που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόληση στην πράξη τη κυρία Οκονή. Ε, εδώ λοιπόν έχει γίνει δουλειά ε, πολύ ε, συστηματική. Γιατί όλοι οι εισηγητέ, οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διερμηνεί του οποίου χαιρετώ, οι νομικέ υπηρεσίε έχουν κάνει όλοι πολύ σκληρή δουλειά. Και δεν έχει τελειώσει η δουλειά αυτή. Πολλοί από εσά και πολλέ από εσά θα επιστρέψετε εδώ και το εύχομαι σε αυτήν την ε, σύνοδο, σε αυτό το σώμα, για να συνεχιστεί το έργο αυτό με τι προτάσει τη κυρία Κράτα, με τι προτάσει τη κυρία Μπόλ. Με τι προτάσει του κυρίου Μπαλντασάρε με τι διαδοτικέ μεταρρυθμίσει τη τράπεζα. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ξέρω ότι τα κείμενα αυτά καθυστέρησαν. Θα ήθελα να τα είχαμε κάνει όλα, όλα τα οριζόντια διατομιακά κείμενα που αφορούν ε, τις 8.300 τράπεζες για τις εγγυήσεις, τις ανακεφαλαιοποιήσεις, το εύρωστο του τομέα αυτού να είχαν έρθει γέρος. Αλλά χρειάστηκε να τα δούμε κατά να τα μελετήσουμε σε κάθε τεχνικό κανόνα. Και με ρωτάνε είναι αρκετά αυτά τα κείμενα για να ρυθμίσουμε τραπεζικό τομέα και απάντησα ναι, ναι, συνολικά αρκούν αρκεί να εφαρμοστούν σωστά. Αλλά είναι αρκετά για τις μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης. Όχι πολλές φορές. Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από της χώρας στην οποία εδράζονται. Δεν αρκεί αυτό και το πρόβλημα δεν είναι απλώς κοινωνικό, είναι συστημικό για ολόκληρη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλησα να υπάρξει αυτή η τελική διαφορετική μεταρρύθμιση και γι' αυτό σωστά θα την εγκρίνει η Σύνοδος της Ολομέλειας και ελπίζω να επανέλθετε στο Κοινοβούλιο, αν το θελήσουν και οι πολίτες, ώστε να προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση. Και εφόσον είμαι και εγώ εδώ θα την παρακολουθήσω στενά γιατί πιστεύω σε αυτήν. Πιστεύω για να διαχωρίσουμε σωστά τη στάθμιση και την διαχείριση του κινδύνου από τα υπόλοιπα. Και ίσως και αυτό που σας πρότεινα, οι κερδοσκοπικές ε, δράσεις και ενέργειες των τραπεζών. Αυτό που ονομάζουμε trading και δεν μπορούν να δικαιολογούνται από την άποψη του κοινού συμφέροντος και τη οικονομία, να διαχωριστούν, να διαχωριστούν για τις μεγάλες, από τις μεγάλες τράπεζες. Ευχαριστώ ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη σωστή υλοποίηση των κειμένων αυτών, να τα να αποτιμούμε, να τα συμπληρώνουμε, να τα διορθώνουμε εφόσον χρειαστεί και να, υπάρχει, να υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού για όλους τους παράγοντες. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γέννησε το G20 όλη αυτή την προσπάθεια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ρύθμισης. Για να μην ξαναυπάρξει τέτοια κρίση. Κάναμε σωστά τη δουλειά μας και θα πρέπει με τους Αμερικανούς κατά κύριο λόγο εταίρους μας αλλά και στα πλαίσια του G20 να βεβαιωνόμαστε ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του στο σπίτι του. Διότι θα ψηφίσετε ένα κείμενο που απεικονίζει τη δουλειά μας κυρίες και κύριοι τραπεζίτε βρίσκουν ότι είναι υπερβολική αυτή η ρύθμιση. Εγώ αυτό που βρίσκω ότι είναι υπερβολικό είναι η απουσία ρύθμιση. Η αυτορύθμιση τη αγορά, την οποία δεν πιστεύω. Είναι η έλλειψη, απόλυτη έλλειψη ρύθμιση. Και αυτοί οι ε, εκτροχιασμοί που βλέπουμε να υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ρύθμιση ε, άνωθεν. Αυτό επιθυμήσαμε και βλέπω κυρία Πρόεδρε ότι όλες οι πολιτικές ομάδες αυτής της ε, Συνόδου έχουν με τον ένα τον άλλο τρόπο συμμετάσχει μέσω των εισηγητών και εισηγητριών που ανέφερα. Δεν είναι η στιγμή να εκφράσουμε την προσωπική μας ικανοποίηση. Είναι εκατομμύρια πολίτες που υποφέρουν, που έχουν δυσκολίες και κάνουν θυσίες για να αντέξουν. Βάσει όμως των όσων ανέφεραν για τη σταθεροποίηση των χρηματαγορών με σωστούς κανόνες θα πρέπει να ενώσουμε όλοι τις προσπάθειές μας για να υπάρχει ανάκαμψη, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ο λόγος των Υπουργό Βενιζέλο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή έτυχε να ασκώ τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών στην Ελλάδα την πιο δύσκολη στιγμή της δημοσιονομικής κρίσης τη στιγμή που η δημοσιονομική κρίση μετατραπόταν και σε κρίση του τραπεζικού συστήματος λόγω και της ανάγκης δραστικής μείωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους μπορώ μέσα από τα βιώματα και την εμπειρία μου να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που γίνεται σήμερα η απόφαση που θα λάβετε σε σχέση με την τραπεζική ένωση σε σχέση με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης είναι μια πολύ σημαντική πράξη τολμώ να πω μια ιστορική πράξη γιατί σπάμε τον δεσμό ανάμεσα στο ενδεχόμενο η δημοσιονομική κρίση να μετατρέπεται σε χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική και το αντίστροφο. αυτόν τον φαύλο κύκλο δεν πρέπει να τον ξαναζήσουμε. η προσπάθεια να συμπληρωθούν τα θεμελιώδη και γενετικά κενά της οικονομικής και νομισματικής ένωσης είναι δύσκολη. η ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης απαιτεί ακόμη πολλές προσπάθειες και συμφωνώ με όσους από τους αξιότιμους βουλευτές τόνισαν προηγουμένως ότι δεν αρκεί να έχουμε έναν μηχανισμό ενιαίο μηχανισμό εποπτείας δεν αρκεί να έχουμε έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης με όσα προβλήματα και ατέλειες έχει χρειαζόμαστε και έναν πραγματικά ενιαίο μηχανισμό προστασίας εγγυήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα ξεπερνά τους στόχους της οδηγίας που είναι στόχοι εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων εγγύησης. αυτό που γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια προσπάθεια να ξεπεραστούν να αρθούν πολύ σημαντικές εσωτερικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών διαρθρωτικές ανισότητες της ενιαίας αγοράς στον χρηματοοικονομικό τομέα. η πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου ανισότητα στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά είναι η ανισότητα των επιτοκίων γιατί αυτή αναπαράγει βαθιές αναπτυξιακές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. όταν μια ελληνική μικρή ή μεσαία επιχείρηση δανείζεται χρήμα από τις τράπεζες με επιτόκιο έξι ή εφτά ακριβότερο από ό,τι δανείζεται μια γερμανική επιχείρηση αναπαράγεται μια εσωτερική αναπτυξιακή και κοινωνική ανισότητα. αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μια τραπεζική ένωση. μια άλλη πολύ σημαντική ανισότητα που αντιμετωπίζουμε ακόμη στην ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι η απόσυρση καταθέσεων για να μεταφερθούν σε άλλη χώρα όχι γιατί υπάρχει καλύτερο επιτόκιο μπορεί το επιτόκιο να είναι μικρότερο αλλά γιατί υπάρχει βαθύτερο αίσθημα ασφάλειας και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. γι' αυτό χρειαζόμαστε και τον τρίτο πυλώνα του ευρωπαϊκού μηχανισμού εγγύησης καταθέσεων για να ξεπεραστούν οριστικά αυτές οι δύο πολύ σημαντικές ανισότητες. υπάρχει τώρα όμως ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. λίγες μέρες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές τώρα που πρέπει όλοι να διατυπώσουμε την ολοκληρωμένη πρότασή μας για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης απευθυνόμενοι σε πολίτες απευθυνόμενη σε νέους ευρωπαίους πολίτες που είναι άνεργοι. το ερώτημα είναι γιατί τους ενδιαφέρει αυτό που γίνεται στην τραπεζική ένωση γιατί είναι σημαντικό για αυτούς να υπάρχει ενιαίος μηχανισμός εποπτείας και ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης καταθέσεων. πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι αυτές είναι προκατακτικές προϋποθέσεις για να στηριχθεί με πιο υγιή και ανταγωνιστικό τρόπο η ευρωπαϊκή πραγματική οικονομία για να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με ίσους όρους με υγιή τρόπο με επιτόκια τα οποία είναι πραγματικά ανταγωνιστικά έτσι αντιμετωπίζουμε το μεγάλο ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη και τελικά η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. έτσι χτυπάμε το πρόβλημα της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων στην καρδιά του. άρα αυτό που γίνεται σε σχέση με την τραπεζική ένωση δεν αφορά τράπεζες τραπεζίτες υβριδικά προϊόντα μετόχους χρηματοοικονομικά παιχνίδια αφορά και αυτό βεβαίως αφορά και αυτή τη σφαίρα την χρηματοοικονομική σφαίρα αφορά όμως εν τέλει και κυρίως την σφαίρα της πραγματικής οικονομίας εκεί που πονά η ευρώπη εκεί που εκφράζει την αγωνία του ο κάθε ευρωπαίος πολίτης και ιδίως αυτός που ζει σε κατάσταση ανεργίας ή οριακά σε κατάσταση πολύ κοντά στη φτώχεια. έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να μιλήσουμε και για όλα όσα πρέπει να γίνουν συμφωνώ με τον επίτροπο τον κύριο μπαρνιέ τον οποίον και εγώ τιμώ και επενώ για τη δουλειά του την αιμονή του τον σταθερό προσανατολισμό του πως πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. σημειώνω ως πολύ σημαντικό βήμα τον απόλυτο διαχωρισμό επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών ως στοιχείο διαφάνειας. έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ποια είναι η αλήθεια σε σχέση με τους στόχους μας στην τραπεζική ένωση. προφανώς και θέλουμε να ελέγξουμε την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των τραπεζών και των επενδυτικών και των εμπορικών. προφανώς και θέλουμε να ελέγξουμε τα κριτήρια και την ποιότητα των δανειοδοτήσεων των χορηγήσεων δανείων εκ μέρους των τραπεζών. Αυτή η έλεγχη μέσα από τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας τελικά βοηθούν στην ανάπτυξη βοηθούν στην υγιή ανταγωνιστικότητα βοηθούν στις επενδύσεις βοηθούν τελικά στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας γιατί πίσω από όλα αυτά υπήρχε η σκέψη πως η χρηματοοικονομική σφαίρα έχει οριστικά αποχωριστεί από την πραγματική οικονομία αυτοτροφοδοτείται πως αποκομίζει εύκολα κέρδη μέσα από χρηματοοικονομικά παιχνίδια και αυτό μπορεί να είναι μια ιστορία χωρίς τέλος ότι έτσι μπορούμε να πηγαίνουμε να πορευόμαστε προς το μέλλον χωρίς κανέναν κίνδυνο σωρεύοντας υπερκέρδη. Ε, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Απεδείχθη ότι δεν οδηγείται πουθενά. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο. Ο έλεγχος της ποιότητας των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, των 130 ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών, τελικά οδηγεί και σε μια έμεση αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων άρα μας φέρνει αντιμέτωπους και με το ζήτημα του ευρωπαϊκού δημοσίου χρέους γιατί φυσικά η διαχείριση του ευρωπαϊκού δημοσίου χρέους του δημοσίου χρέους των κρατών μελών δεν μπορεί να γίνει μόνο από τα κράτη ή την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας. χρειαζόμαστε το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αλλά χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα που είναι βέβαιο πως Μετέχοντα στην αγορά κρατικών ομολόγων στην ευρώπη αποκτά και διατηρεί ένα υγιές χαρτοφυλάκιο το οποίο με τη σειρά του βοηθάει τις πραγματικές οικονομίες των κρατών μελών. έτσι μπορούμε να περάσουμε από την εμπειρία του φαύλου κύκλου σε έναν κύκλο εξυγίανσης ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε στους ευρωπαίους πολίτες μιλώντας τους για πράγματα που τους αφορούν εξηγώντας τους ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι αφηρημένα δεν αφορούν ένα κλειστό κόσμο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών αλλά αφορούν την πραγματική ευρώπη τις ευρωπαϊκές κοινωνίες τους λαούς και τους πολίτες. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ο λόγος στον κύριο Χέκμαρκ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Μπαρνιέ, τον κύριο Βενιζέλο, την Ελληνική Προεδρία και την προηγούμενη, τη Λιθουανική, που μας επέτρεψε να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και τώρα είμαστε στην τελική περίοδο εντατικών νομοθετημάτων όπου θέσαμε τα θεμέλια για το μέλλον του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και της τραπεζικής νομοθεσίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία εδώ μεταξύ των δημοσίων οικονομικών και της ε, ε, εξασφάλισης της οικονομίας γενικότερα και μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο όπου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η σταθερότητα θα συμβάλλει και εκείνη στις επενδύσεις και την απασχόληση που χρειαζόμαστε. Τώρα δημιουργούμε τα θεμέλια ενός τραπεζικού τομέα σταθερότερου με τη διαδικασία διάσωσης με ίδια μέσα που συζητήσαμε πιο πριν για να έχουμε πιο πολύ σταθερότητα στο σύστημα ε, όταν έρθει η επόμενη κρίση. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε κοινή νομοθεσία και ανάληψη ευθυνών σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να είμαστε πιο αξιόπιστοι να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη που χρειάζεται η Ευρώπη. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι, οι φορολογούμενοι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα. Όταν επενδύει κανείς σε τράπεζες θα πρέπει να αναλαμβάνει τον κίνδυνο τον επιχειρηματικό όπως και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Θα πρέπει να, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε το ε, συνολικό σύστημα. Τώρα έχουμε μια δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Ευχαριστώ όλους τους συμμετασχόντες στη συζήτηση για την ευρεία υποστήριξη του μέτρου. Τώρα πρέπει να φροντίσουμε για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων και τέλος να έχουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση που χρειάζεται τόσο πολύ η Ευρώπη. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια και ε, περηφανεύομαι που συμμετείχα και εγώ σε αυτά, σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Χόκμαρκ. Για δύο λεπτά κύριο Σίμων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Επίτροπε Παρνιέ, αξιότιμε Υπουργέ, κύριε Βενιζέλο, αγαπητοί συνεισηγητές, ε, σκιώδεις εισηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που μετά από πέντε χρόνια συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση να μπορούμε να κλείσουμε πλέον το θέμα αυτό. Στην αρχή της συζήτησης παρουσιάστηκε η θέση των, της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας. Στόχος μου είναι στο τέλος της συζήτησης να περάσω, να στείλω ένα μήνυμα από το κοινοβούλιο αυτό προς όλη την Ευρώπη. Ότι κάναμε δηλαδή ένα σημαντικό βήμα που θα το ολοκληρώσουμε αργότερα στην ψηφοφορία. Παρά τις κριτικές φωνές ε, που ε, παρά τις κριτικές ε, φωνές ε, που μας επετέθησαν, παρά τις φωνές όλων εκείνων που δεν πίστευαν στο προοπτική της επιτυχίας, τα καταφέραμε. Τώρα, όπως είπα και πιο πριν, οι φορολογούμενοι δεν είναι πια στην πρώτη γραμμή του πυρός, αλλά μετατίθενται στα μετόπισθεν και στις μελλοντικές κρίσεις που θα υπάρξουν ε, θα έχουμε ε, ελεγχόμενες διαδικασίες από ό,τι κατά το παρελθόν. Εμείς κάναμε τη δουλειά που μας αναλογούσε. Πολλά μέλουν να γίνουν και στην επόμενη θητεία και βεβαίως ε, οι επόμενες γενναίες, οι διάδοχοι της Επιτροπής πολλά έχουν ακόμα να κάνουν. Αλλά το μήνυμα για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι σημαντικό. Η Ευρώπη απέδειξε άλλη μια φορά ιδιαίτερα σε περιόδους βαθιάς κρίσης είναι σε θέση να ε, εξέρχεται ενισχυμένη και πρέπει να πούμε ότι και οι κρίσεις συνέβαλαν στην πρόοδο της Ευρώπης και η χρηματοοικονομική ε, και οικονομική κρίση ε, έδωσε κάποια θετικά στοιχεία. Τώρα ε, μπορούμε να μιλήσουμε για εξασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας για τους πολίτες. Βαδίζουμε προς τα μπρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σίμων. Κλείνει η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι κοινή συζήτηση για την ασφάλεια των προϊόντων και προστασία των καταναλωτών. Τρεις εκθέσεις έχουμε. Της κυρίας Σάλντεμόζα, της κυρίας Πίτικάινεν